bitte Platz zu nehmen. Παρακαλώ, καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ich möchte den nächsten Θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το οποίο προβλέπει ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση με τον κύριο Κρόισμαν. πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης μέχρι την εκλογή της Βουλής και νυν πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας που είναι η Βερκόφνα Ράντα. Και όταν ε, υπηρετούσε την κυβέρνηση απεδείχθη ένθερμος υποστηρικτής ε, της μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία, τις οποίες και προώθησε. Και οι πρωτοβουλίες αυτές σήμερα είναι σημαντικότερες από ποτέ, γιατί θα πρέπει η Ουκρανία να γίνει υπόδειγμα προς μίμηση, ε, να επιτύχει τουλάχιστον εκείνη που δεν είναι υπορωσική κατοχή ε, εκείνο το κομμάτι και με την βοήθειά μας και την οικονομική και την τεχνική γιατί είναι αλληλένδετα αυτά ε, θα πρέπει να προχωρήσουν τα έργα και οι μεταρρυθμίσεις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Και ξέρετε τον Οκτώβριο έχουν δημοτικές εκλογές ήδη κοντά. Και θα πρέπει κάπως να έχει ιδρυωθεί η γραμμή μας και να έχουμε και ιστορίες επιτυχίες, ε, success stories, στη διαδικασία μετασχηματισμού σε κράτος δικαίου, σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάποια οικονομική τάξη. Στο Στρασβούργο, κύριε Πρόεδρε, τον Ιανουάριο, ε, ψηφίσαμε ε, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία ένα πάρα πολύ σημαντικό και σαφέστατο ψήφισμα. Τις περασμένες ημέρες το τονίσαμε και σήμερα ψηφίσαμε την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εξωτερική δηλαδή και πολιτική ασφαλείας και πάλι διατρανώνουμε αυτή τη θέση ότι η Ουκρανία είναι θύμα ε, έξωθεν εισβολής, έχει παραβιαστεί το διεθνές δίκαιο οι αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας των λαών επίσης και η Ρωσία φέρει εδώ την ευθύνη όχι ως σιωπηρός παρατηρητής αλλά ως εμπλεκόμενο και εμπόλεμο μέρος και ως ε, εμπλεκόμενο μέρος φέρει και ευθύνη για την ειρήνευση και κυρίως για την υλοποίηση και εφαρμογή της Συμφωνίας του Μίνσκ. Είναι συντριπτική πλειονότητα του κοινοβουλίου σε αυτή τη γραμμή και την εκπροσωπώ λέγοντας αυτά. Θέλω να σας δώσω αμέσω το λόγο που ήρθατε εδώ και θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τους συναδέλφους και με δική μας αντιπροσωπεία για να έχουμε στενή συνεργασία στην Ουκρανία. Βλέπω μόλις τον πρόεδρο, συνάδελφο Πλένκοβιτς που είναι πρόεδρος αντιπροσωπεία με την Ουκρανία, ο οποίο και θα με αντικαταστήσει αμέσω στην Προεδρία διότι πρέπει να είμαι στο Βερολίνο απόψε και πρέπει να βγάλω και ένα λόγο ακριβώ για αυτό το θέμα και θα αναγκαστώ να αποχωρήσω. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι από την Ουκρανία, καταρχάς κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη θέση σας όσον αφορά στην Ουκρανία, αλλά και για τη στήριξή σας. και καλό να είναι να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η αξιολόγησή σας είναι πολύ αντικειμενική για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Η χώρα μας υποφέρει από τη ρωσική κατοχή και οφείλουμε να το πούμε αυτό και να αποκαλέσουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είναι μόνο μια επίθεση στο ουκρανικό έδαφος, είναι μια επίθεση και στις ευρωπαϊκές αξίες, τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Όλα αυτά χρειάζονται την κατάλληλη δράση, την αντίστοιχη δράση από πλευράς υπολείπου κόσμου. Για μένα λοιπόν αυτή η δήλωση είναι, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Σήμερα πριν από ένα χρόνο στις παραμονές της επανάστασης της αξιοπρέπειας και της επονίδης της διαφυγής του τότε Προέδρου της Ουκρανίας, η ΕΕ και το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό αναγνώρισαν τη Βερκόβνα Ράντα ως το μόνο ε, νόμιμο όργανο ε, κυριαρχίας. Το Κοινοβούλιο ανέλαβε την αποστολή να αποκαταστήσει την τάξη στη χώρα και να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες του ουκρανικού λαού για ένα ευρωπαϊκό δημοκρατικό κράτος. Να γίνει η χώρα μας μέρος του ευρωπαϊκού ε, ε, σπιτιού, αν θέλετε, της ευρωπαϊκής οικογένειας. Το τελευταίο χρόνο, λοιπόν, έχει αποκατασταθεί το σύστημα διακυβέρνησης, υπάρχει νέος πρόεδρος, έχει εκλεγεί κοινοβούλιο, έχει υπογράψει η Ουκρανία η Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΕ. Σήμερα λοιπόν με την πρώτη μου επίσκεψη στο εξωτερικό ως πρόεδρος του Ουκρανικού Κοινοβουλίου μαζί με τον πρόεδρο Σούλτς θα ε, κηρύσουμε την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης της, ε, κοινοβουλευτικής, της Επιτροπής Σύνδεσης Κοινοβουλίων. Αυτό είναι σημαντικό εργαλείο για να υλοποιήσουμε την ιστορική συμφωνία. Δύο είναι οι προκλήσεις. Πρώτον να υπερασπιστούμε τις ευρωπαϊκές αξίες ελευθερίας δημοκρατίας, να σταματήσουμε την εξωτερική επίθεση, να διατηρήσουμε την εδαφική ακαιρεότητα και εθνική κυριαρχία και να εδραιώσουμε την Δεύτερον, να έχουμε θεσμική μεταρρύθμιση για, έτσι ώστε μια μετασοβιετική δημοκρατία να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Το, δεν είναι εύκολο από τη μία να είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και από την άλλη να υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις. Έχουμε όμως ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις. Έχουμε τη στρατηγική για την εθνική ανάπτυξη με ορίζοντα το 2020. Η συμφωνία υλοποίησης της συμφωνίας, το σχέδιο υλοποίησης της συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΕ είναι σημαντικό, αλλά και η συμφωνία ε, συμμαχίας της κοινοβουλευτικής ε, πλειοψηφίας. Έχω ξεκινήσει με βάση όλα αυτά τα κείμενα μια διαδικασία κατάρτιση σχεδίου νομοθετικής στήριξης των μεταρρυθμίσεων για τη διετία 15-17. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει αυτό το σχέδιο στο Κίεβο και θα τεθεί προς διαβούλευση στα υπόψη των μελών του Κοινοβουλίου, του Προέδρου και της Κυβέρνησης. Με αυτή τη δουλειά για το σχέδιο στήριξης των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας θα γίνει και η λοκομοτίβα για συστημικές μεταρρυθμίσεις, για να τηρήσει η Ουκρανία τις εγχώριες και διεθνείς της δεσμεύσεις. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο μας να είναι το εργοστάσιο παραγωγής της ε, μεταρρυθμιστικής νομοθεσίας. Τι όμως έχει ήδη γίνει. Χάρη στις κοινέ προσπάθειες ε, ε, Κοινοβουλίου Προέδρου και Κυβέρνησης της Ουκρανίας ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε το ένα νομοθετικό πακέτο κατά τη διαφθοράς. Από τον περασμένο Οκτώβριο υιοθετήσαμε διάφορους νόμους για να στηρίξουμε τις δράσεις του Εθνικού Γραφείου κατά τη διαφθορά γιατί η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ουκρανίας. Πρέπει να το σταματήσουμε, να εξαλείψουμε, να ξεριζώσουμε αυτό το φαινόμενο της διαφθοράς ε, στη χώρα μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε ε, τη θέση του Διευθυντή σε αυτό το γραφείο μετά από μια διαφανή διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Και Έχουμε ε, συμφωνία, έχουν γίνει βήματα για τη μεταρρύθμιση του, της δικαιοσύνης, ε, έχουμε νομοθεσία για το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη και έχουμε υιοθετήσει μια σειρά από νομοθετήματα για να ενισχύσουμε την αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας. Ως προς την αποκέντρωση τώρα και τη συνταγματική μεταρρύθμιση, είναι μια δουλειά που προχωράει, είναι πολύ σημαντική, είναι, μια από, είναι ένας από τους κλάδους πρώτης προτεραιότητας ε, για τη μεταρρύθμιση στην Ουκρανία Πρέπει να έχουμε ένα ποιοτικό επίπεδο διακυβέρνηση. αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, το σύστημά μας πρέπει να έχει ποιότητα. Έχουμε ήδη λάβει αποφάσεις για την ε, φορολογική αποκέντρωση ή τη δημοσιονομική αποκέντρωση και έχουμε θετήσει νόμου για περιφερειακή πολιτική και για την εθελούσια σύνδεση των κοινοτήτων. Ε, η επιτυχία της διαδικασίας αποκέντρωσης και όλων των μεταρρυθμίσεων θα εξαρτηθεί από τη βελτίωση του συντάγματος. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει ξεκινήσει τη σύσταση μιας επιτροπής που μαζί με ε, επιτροπή σοφών, με εμπειρογνώμων, με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών θα προετοιμάσει τις ε, προτινόμενες αλλαγές στο ε, Σύνταγμα. Και σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος έχουμε επιτέλους την ευκαιρία να εγκρίνουμε σχετική νομοθεσία στις αρχές ε, Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις προτάσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Θέλω να τονίσω ότι ε, ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες συνταγματικής μεταρρύθμισης και αποκέντρωσης πριν από τη διαδικασία του Μίνσκ και σας διαβεβαίω οι περιφέρειες της Ουκρανίας θα έχουν εξουσίες και αυτό θα είναι απότοκο των μεταρρυθμίσεων και έτσι θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όλων όσοι ουσιαστικά και με ειλικρίνεια θέλουν την αλλαγή και δεν επινοούν τεχνάσματα για να κρύψουν τις διεκδικήσεις τους για την εξουσία ε, θα έχουμε ένα σύστημα αποκέντρωσης μεταρρυθμίσεων και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι ε, η οικονομική επιτυχία της Ουκρανίας αυτή είναι, θα είναι τελικά και η πιο επιτυχημένη κύρωση έναντι της ρωσικής ε, πολιτικής. Χωρίς ε, διεθνή βοήθεια είναι αδύνατο να σταθεροποιηθεί η Ουκρανική οικονομία και θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικές συζητήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε το τρίτο πρόγραμμα μακροοικονομικής βοήθειας. Η Ουκρανία μεταρρυθμίζεται ε, κάτω από τους ήχους των κανονιών και δίνει πάρα πολύ, πολλούς και σημαντικούς οικονομικούς και πολιτικούς πόρους προκειμένου να αφαιρεθεί σε αυτόν τον αγώνα να αποτρέψει τον επιτιθέμενο. Η Ρωσία ε, παρόλο που είναι συμβαλόμενο μέρος στο μνημόνιο της Βουδαπέστης και έχει δεσμευτεί ότι θα απέχει από την απειλή τη χρήση της ε, βίας ε, έναντι της πολιτικής ανεξαρτησίας της Ουκρανίας και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα όπλα της εναντίον της Ουκρανίας συνεχίζει τις επιθέσεις και παρά τις συμφωνίες του Μίνσκ οι Ουκρανοί συνεχίζουν να βρίσκουν το θάνατο καθώς τον ε, χρόνο πύραυλοι της Ρωσίας ε, ουσιαστικά δημιουργούν θρήνο και τεράστια οδύνη στις οικογένειες των Ουκρανών σε όλη την χώρα. Πάνω από 5.000 Ουκρανοί έχουν βρει το θάνατο από, τη, από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις στον Ντόνμπας. Παράλληλα, ο αριθμό των εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων αυξάνεται, έχει φτάσει στο 1 εκατομμύριο και οφείλουμε ευγνωμοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί χάρη σε πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου υπήρξε ψήφισμα τον περασμένο ε, Ιανουάριο και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο, σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ρωσία συνεχίζει να στηρίζει την τρομοκρατία, τι τρομοκρατικέ επιθέσει, αρνείται τη στρατιωτική τη παρουσία στην Ουκρανία, ενώ αυτή είναι πρόφα Νης. Τα γεγονότα στον Τελμπάτσεβο την περασμένη εβδομάδα δείχνουν τον τακτικισμό τη Ρωσία. Σχέδιο του Κρεμλίνου είναι να καταλάβει την πόλη πριν την εκεχηρία στι 15 Φεβρουαρίου. Οι τρομοκράτε αγνώρισαν τι συμφωνίε του ΜΙΣ και συνέχισαν τι επιθέσει του και κατάκαψαν την πόλη. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας και Άμυνα τη Ουκρανίας αποφάσισε να προσφύγει στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πρόταση να, αποστολή, να αποσταλεί ε, να να οργανωθεί μια αποστολή διατήρησης της ειρήνης στην Ουκρανία. Ε, διανικό θα ήταν να είναι αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ε, θα πρέπει να πούμε ότι το σφράγισμα των συνόρων και η παρακολούθηση από τον ΑΣΕ και από τους παρατηρητές που είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ειρήνης, αυτό θα μπορέσει να εκθέσει την παρουσία ε, ρωσικών στρατευμάτων. Θα αναγκάσει τη Ρωσία να αποτραβηχθεί από την Ουκρανία, να αποσυρθεί. Συνεχίζει η Ρωσική Ομοσπονδία να χειραγωγεί τις εξελίξεις και παρόλο που η στάση της Ουκρανίας είναι ειλικρινής, χρησιμοποιούνται οι συμφωνίες του Μίνσκ ως προ πέτασμα καπνού πίσω από πράξεις που μόνο στόχο έχουν να καταστρέψουν την Ουκρανική ανεξαρτησία, ελευθερία και δημοκρατία. Ε, οι Ουκρανοί πολίτες ε, κρατούνται παρανόμως σε ρωσικό έδαφος, π.χ. μέλος του Ουκρανικού Κοινοβουλίου, η κυρία Ναντίγια Σαυτσέγκο η οποία ε, ε, κάνει απεργία πείνα σε 74 μέρες τώρα. Ευχαριστώ τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργή δράση που έχουν υιοθετήσει για τις πρωτοβουλίες τους υπέρ της απελευθέρωσής της. Σας καλώ και σας απευθύνω έκκληση να μην σταματήσετε. Η αυξημένη πίεση στη Ρωσία από τη διεθνή κοινότητα θα την εξαναγκάσει να σταματήσει τις επιθέσεις. Αγαπητοί φίλοι, θέλω να υπογραμμίσω τη σαφή θέση της Ουκρανίας. Δεν βλέπουμε εναλλακτική ε, λύση ε, παρά μόνο μια ειρηνική επίλυση του προβλήματος. Ε, το να λυθεί το πρόβλημα εξαρτάται κατά βάση από τη ρωσική πλευρά, η οποία έχει σπαταλήσει πάρα πολλές ευκαιρίες να αποδείξει τη δέσμευσή της στην ειρήνη, με πράξεις και όχι με λόγια. Θα πρέπει η Ρωσία να μπει σε έναν ειλικρινή ε, διάλογο και για να γίνει αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς κυρώσεων, να ενισχυθούν τα περιοριστικά μέτρα σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, να συνεχιστεί διπλωματική και πολιτική πίεση ε, στο Κρεμλίνο και να έχει η Ουκρανία ουσιαστική βοήθεια και στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Είναι πήγον να βελτιώσουμε τις αμυντικές ικανότητες της Ουκρανίας και να έχει η Ουκρανία έξυπνα αμυντικά όπλα για να αμυνθεί στο ουκρανικό έδαφος από τις ρωσικές επιθέσεις. Μόνο τότε θα καταλάβει το, κρε... το Κρεμλίνο ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να αντιταχθεί στη ρωσική επίθεση. Και ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξει αυτή την προσέγγιση. Και σας καλώ να θυμηθείτε και το θέμα της Κρυμαίας. Ένας χρόνος θα έχει περάσει πολύ σύντομα από την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ένας χρόνος οικονομικής υποβάθμισης και ε, ε, καταστρατηγήσεων των δικαιωμάτων των, πληθυσμών Τατάρων ε, και Ουκρανών της Κρυμαίας. Η Ουκρανία θα ήθελε να αναθεωρηθεί συνολικά το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της ε, Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο και να υιοθετηθεί σχετικό ψήφισμα. Ε, σας απευθύνω έκκληση να συνεχίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχολείται με το θέμα της Ουκρανίας εσείς παρακινείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση να, έχει πιο να παρέχει πιο αποφασιστική στήριξη στην Ουκρανία. Εσείς διαμορφώνετε την κοινή γνώμη στην Ευρώπη. Εσείς αντιστάσεστε στην ρωσική ε, προπαγάνδα. Όλα αυτά είναι πράγματα που περιμένει η Ουκρανική ε, κοινωνία. Περιμένουμε ότι ε, την παραμονή της Συνόδου για την ε, εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ανατολά στη Ρήγα, το Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα ενθαρρύνουν το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στείλει ισχυρό πολιτικό μήνυμα, να αναγνωρίσει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας μας, να υπάρξει πολιτική απόφαση για ένα καθεστώς ε, χωρίς θεωρήσεις για σύντομα ταξίδια Ουκρανών πολιτών. Είναι κάτι που αξίζουν οι Ουκρανοί πολίτες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμότατα και ειλικρινέστατα για την παρουσίαση αυτή. 16 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο και θα επιθυμούσα εδώ να κλείσουμε τον κατάλογο και με την άδειά σας να πω ότι ε, ο χρόνος αγόρευσης είναι το πολύ 1,5 λεπτό. Συμφωνείτε? Μάλιστα. Ο συνάδελφος παρακαλώ να αναλάβει και την Προεδρία. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Μπρόκ, κύριε Πρόεδρε Γκρόισμαν, κύριε Πρεσβευτά και καλώς ορίζω και τους βουλευτές από το Εκκληνικό Κοινοβούλιο. Από ό,τι βλέπω ότι ο πρόεδρος Γκρόσμαν με βαλέει παριθμόν ένα ε, υπό την ιδιότητα του επικεφαλής ε, για την αντιπροσωπεία με την Ουκρανία και θέλω να πω ότι μετά τη συνεδρίαση αυτή θα έχουμε την αναρκτήρια σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης και χαιρετίζω εδώ και τον κύριο Σέμερα και τον ομολογό μου που είναι εδώ και θα συζητήσουμε ένα ολόκληρο κατάλογο για θέματα ανθρωπιστικά, θέματα ασφαλείας, πολιτικά θέματα, κυρίως στην Ανατολική Ουκρανία και αύριο την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης, πολιτικά, οικονομικά, ενεργειακά θέματα. Ανυπομονώ για τη συζήτηση αυτή. Όπως είπατε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί τα μάλα για την Ουκρανία με αρκετά ψηφίσματα, πολλοί βουλευτές ε, θέλουν να σας βοηθήσουν σε αυτές τις δύσκολες ε, στιγμές όπου δέχεστε επίθεση. Θα θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτή τη στήριξη και την ισχυρή δέσμευση. Και για να μην μακρηγορήσω θα σας ζητούσα να μας εξηγήσετε στις απαντήσεις σας Πώς ε, βλέπετε περαιτέρω διεθνείς δεσμεύσεις ε, για ε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ολοκλήρωση με την Ουκρανία των σημερινών εδάφων που είναι κατοχή Ίσως θα θέλαμε και κάποια περαιτέρω διευκρίνηση των ιδεών. Ακούσαμε και τον κύριο Προσέγκο και τον πρόεδρο του ΕΣΕ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο, στην κυρία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Γκρόσμαν, καλώς ορίσατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συνεχίσω στα λετωνικά γιατί αυτή είναι ε, η πρώτη φορά που έχουμε την Προεδρία στο Συμβούλιο. Κυρίες και κύριοι, πριν ένα χρόνο στις 20 Φεβρουαρίου επισκέφτηκα το Κίεβο και ήμουν στην Βερχόβνα Ράντα όπου συναντήθηκαν ε, διάφορες βουλευτές για να πάρουν μια ιστορική απόφαση να αποτρέψουν περαιτέρω βία. Ήμουν εκεί και είδα θύματα ε, βίας, ε, ανθρώπους που είχαν υποστεί επιθέσεις. Εγώ Βέβαια ότι μόνο αν η Ουκρανία μπορέσει να προστατεύσει τον εαυτό της θα έχουμε μια αίσια έκβαση και θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να βοηθήσουν την Ουκρανία να ενδυναμώσει την αμυντική της ικανότητα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, προχωρούν οι διαπραγματεύσεις σε σχέση με την ανάπτυξη της ερνευτικής δύναμης ε, του ΟΗΕ στην Ουκρανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σάντρα. Η κυρία Γκόμες, παρακαλώ. Κύριε Γκρόσμαν, καλωσορίσατε. Στις 21 Φεβρουαρίου πέρσι ήμουν στο Ευρωμαϊντάν και την επόμενη μέρα ξυπνήσα και είδα ότι ο Γιαννούκοβιτς ε, είχε φύγει. Και μαζί με άλλους συναδέλφους που έφτασαν το μεταξύ είδαμε την ε, φανταστική συμπεριφορά του λαού της Ουκρανίας. Αλλά ταυτόχρονα ανέμεναν ότι θα έρχονταν οι μπελάδες και τώρα έχουν έρθει αυτοί οι μπελάδες και δεν ε, αφορά μόνο την Ουκρανία, μας κλείτει όλους την Ευρώπη και την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας και πρόκειται και για το τι είμαστε. Είμαστε παλιά Ευρώπη, που έχει να κάνει με την παλιά Ρωσία ή αν, είχαμε, ή είμαστε μια νέα Ευρώπη διαρθρωμένη, στενισμένη. Έρχομαι από την Πορτογαλία, δεν ε, είμαι κοντά στα σύνορά σα. αν ε, και πραγματικά ε, τρέφουμε πολύ μεγάλη συμπάθεια, γιατί έχουμε και σημαντική ουκρανική κοινότητα στη χώρα μας, αλλά γιατί καταλαβαίνουμε ότι εδώ πρόκειται για μας, όχι απλώς για σας, για το τι είμαστε και το τι περισπιζόμαστε. Και επομένως συμφωνώ μαζί σας ότι πιθανότατα πέρα από την υποστήριξη που θα έπρεπε να πάρετε και εντός και εκτός Ευρώπης, τίποτα δεν θα είναι πιο σημαντικό από τα όνα ε, αντισταθείτε στην επίθεση του κυρίου Πούτιν και να προχωρήσετε προς την οικοδόμηση δημοκρατίας και την σταθεροποίηση στην Ουκρανία τίποτα ε, δεν θα είναι πιο σημαντικό παρά να ιτηθεί αυτή η επίθεση που υλοποιεί ο κύριος Πούτιν ε, απέναντί σας και απέναντι όλων μας, γιατί τώρα κατανοώ ότι έχουμε ε, και μια απειλή σε όλες μας τις Ευρώπης ότι αφορά τις στρατιωτικές πτήσεις που δεν είναι αναγνωρισμένες. Ευχαριστώ την κυρία Γκόμες, ο κύριος Τόνε, Τάνο, από Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω από την ομάδα του ECR και θα ήθελα να σας πω ότι εμείς κάναμε έκκληση να απελευθερωθεί η κυρία Σαφτσένσκο, την οποία πήγαν οι Ρώσοι σε ουκρανικό έδαφος. Και φυσικά μας δείχνει αυτό ότι είναι ενεργοί και παρόντες. Το 2002 έγραψε ένα άρθρο στη Wall Street Journal που παρουσίασε την ευρωπαϊκή προοπτική ε, για την Ουκρανία. Τότε κανείς δεν θεωρούσε ότι αυτή ήταν και μια πιθανή, μια δυνατή έννοια. Ε, και τότε είχαμε την πορτοκαλία Επανάσταση. Ε, όμως τότε κανένας δεν έδινε τη δυνατότητα ουσιαστικά να εισβάλλει η Ρωσία στην Ουκρανία. Όμως πρέπει να δούμε δούμε τι λέει ο Πούτιν εδώ και 10 χρόνια και ποτέ δεν έκρυβε τις φιλοδοξίες του να δημιουργήσει και πάλι ε, μια μεγαλύτερη αυταρχική Ρωσία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε γιατί υποψιάζομαι ότι η Συμφωνία Μίνσκ 2 δεν θα κρατήσει, δεν θα τηρηθεί. Απλώς εξαγοράζουν χρόνο οι Ρώσοι πριν να προχωρήσουν περαιτέρω προς τη Μαριούπολη ή πριν να δημιουργήσουν ένα χερσαίο διάδρομο προς την Κρυμαία. Υποστηρίζω όλες τις προσπάθειες του Διεθνούς Δημοτικού Ταμείου, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταθεροποίηση της οικονομίας σας, αλλά τι μπορεί να γίνει ε, σε σχέση με το να ε, αποκτήσουν ε, οι δυνάμεις στα μέσα για να αυτοπροστατευτούν, να αυτοεμεινθούν. Υπάρχει δυνατότητα σταθεροποίησης και πώς εξελογείται την έκθεση των New York Times Κάποιοι που ήταν ε, υπεύθυνοι για τη βομβιστική επάθεση μπορεί να έχουν ε, εκπαιδευτεί από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, στην SPU, στο να κατασκευάζουν βόμβες. Ε, και υπάρχει δυνατότητα και GB να προβεί σε κάποιες επιθέσεις βομβιστικές. Αναφέρομαι στην επίθεση στο Κάρκιβ Ευχαριστώ, Τσάρλ. Θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι έχουν ένα μισή λεπτό για να μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο σε αυτή την ειδική περίσταση. Ο κύριος Βαν Ευχαριστώ. Καταρχήν, κύριε Γκρόσμαν, σας υποστηρίζουν ένθερμα οι φιλελεύθεροι σε αυτό το κοινοβουλίο γιατί ε, το ε, έχει ένα παράδειγμα για τις ελεύθερες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές και το Euromaidan είναι ένα παράδειγμα, ένα μοντέλο που θέλει να αποφύγει ο Πούτιν. Δεν θέλει ε, μια ευρωκόκκινη πλατεία ο Πούτιν γιατί αυτό θα τέλο τέλος στην κρίση και στην επίθεση και ακριβώ αυτό δεν θέλει ο Πούτιν πέρα από τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ε, να ε, καταστήσει τους γείτονες τους ε, ανάπηρους. είπατε ότι θέλετε να φέρετε αλλαγές στην Ουκρανία και ότι αγωνίζεστε ως Κοινοβούλιο για την επιβολή μεταρρυθμίσεων, γιατί πρέπει να υπάρχει κράτος δικαίου, πρέπει να υπάρχουν οικονομικές μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις στο στρατό, καταπολέμηση της διαφθοράς και αυτά μπορούν να γίνουν μόνο από ένα ισχυρό κοινοβούλιο και ένα ισχυρό κοινοβούλιο έχει εκλεγεί. Επίσης είμαι περήφανος που από αυτό το κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Έχουμε μια ισχυρή αντιπροσωπεία που συνεργάζεται με τη Ράντα. Έχουμε μια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ε, και έχουμε και μια κοινοβουλευτική ομάδα, πρόεδρος ο οποίος είναι ο κύριος ε, Αουστρεβίξους. Θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία γιατί τη χρειάζεστε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοχμπίλαρ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε της Βολής. Στην αρχή της ομιλίας σας εξηγήσατε ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες ε, δρομολογείται αυτό τον καιρό. Θα ήθελα να δανειστώ μία την ενδεχόμενη κύρωση του ε, ε, Διεθνούς Δικαστηρίου ποινικού δικαστηρίου θα ήταν πολύ καλό για την Ουκρανία πραγματικά αν εργαστείτε προς τη αυτή. Από το 2003 το έχω κοιτάξει οι βουλευτές του Κοινοβουλίου σας εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή και θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, η άποψή σας. Υπάρχει τώρα δυνατότητα να εντατικοποιηθεί αυτή η διαδικασία κύρωσης του καθεστώτο τη Ρώμη για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και δεύτερο, θα χαιρόμουν πάρα πολύ να μας υποστηρίξετε, γιατί υπάρχει μια πρωτοβουλία βουλευτών παγκοσμίω, Parliamentarians for Global Actions, και το Μάρτιο θα γίνει σχετική εκδήλωση στο δικό σα κοινοβούλιο για να ζητηθεί η κύρωση αυτή και θα χαιρόμασταν πάρα πολύ αν μπορούσατε και εσείς από την πλευρά να υποστηρίξετε την εκδήλωσή μας. Ευχαριστώ κυρία Λοχμπίλε και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Σαφχάουζερ, παρακαλώ. Κύριε Πρέσβη, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω την επιθυμία σας να κάνετε. Ε, ο πρόεδρος διορθώνει, τον αποκαλείται κύριε πρόεδρο, όχι κύριε πρέσβη. Λέω λοιπόν ότι ε, χαίρομαι για τα όσα εξαγγέλλεται, αλλά Ας μην γελιέστε. Αυτά τα πολεμοχαρή που ακούτε εδώ στο Κοινοβούλιο δεν είναι ο λόγος της Γαλλίας, ούτε της Γερμανίας, ούτε της Αγγλίας, ούτε των παρατηρητών του ΟΣΕ. Δεν μιλούν για ρωσική κατοχή. Το κοινοβούλιο εδώ λοιπόν είναι απομονωμένο στην εξτρεμιστική του ανάλυση από την κατάσταση γιατί οθείται από ορισμένου θερμοκέφαλους πόλεμοχαρείς που σε καμία περίπτωση δεν εκπροσωπούν τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη. Εδώ το Κοινοβούλιο εργάζεται κατά της Ευρώπη και κατά των ευρωπαϊκών κρατών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Μίνσκ. Θα ήθελα να σας κάνω μία και μόνη ερώτηση κύριε Πρέσβη που ανέκαθεν ήταν δική μου άποψη. Το Μίνσκ 2 έχει το πλεονέκτημα ότι επανακαθορίζει ότι η Ρωσία σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητεί τα σύνορα της Ουκρανίας, τα σημερινά. Διότι επαναλαμβάνει και ξεκαθαρίζει ότι... Αγαπητέ μου συνάδελφοι, σας παρακαλώ, αφήστε με να μιλήσω. Και εγώ σας ακούω στη ιδεολογία σας. Ε, ορίζεται λοιπόν εκεί στο Μίνσκ 2 ότι όταν γίνουν δημοτικές εκλογές, πράγμα που εσείς εγκρίνατε, ε, θα ανακτήσετε στα σύνορά σας την πλήρη σας κυριαρχία. Έρχομαι λοιπόν τώρα να σας ρωτήσω το εξής. Λέγω, πώς θέλετε να διοργανώσετε δημοτικές εκλογές και το καθεστώς αυτονομίας των ανατολικών περιφερειών. Σας ευχαριστώ εξοχότατε κύριε Πρέσβη για να μείνουν όλα πέντα κάθαρα ως προς το ρόλο της Ρωσίας. Ευχαριστώ κύριε Σαφχάουζε. Ίσως έχει σημασία να γνωρίζετε ότι ο κύριος Γκρόισμαν είναι πρόεδρος της Βουλής της Ουκρανίας και δεν είναι πρέσβης, έτσι, προς ενημέρωσή σας. Ε, θα δώσω αμέσως το λόγο τώρα στον κύριο Στέτινα. Παρακαλώ, έχετε λόγο. Ευχαριστώ. Δεν έχετε πια το λόγο, το έχει κύριο Στέτινα. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα ήθελα να πω στον συνάδελφο από τη Γαλλία ότι θέλω και εγώ να μιλήσω και αν έχει την καλοσύνη να με αφήσει να το κάνω. Ε, κύριε Στέτινα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έλεγα ότι θέλω να πω στον Γάλλο συνάδελφο ότι τον παρακαλώ να με ακούσει και εμένα και να με αφήσει να μιλήσω για την σειρά μου. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, αξιότιμο κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να πω το εξή. Τιμώ πάρα πολύ τους μαχητές ε, των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων αλλά και των εθελοντών. Η Ουκρανία ε, δεν έχει αγωνιστεί και δεν αγωνίζεται μόνο για τη δική της ανεξαρτησία αλλά και για την Ευρώπη και γενικότερα τις ευρωατλαντικές αξίες. Εξού και ευγνωμονώ πάρα πολύ τους Ουκρανούς και θαυμάζω τον αγώνα σας. Έχω πάει ε, στον Ντομπάς πρόσφατα και στην περιοχή που έχουν υποτίθεται απελευθερώσει ε, ε, οι αντάρτες. Ε, όλοι οι εκπρόσωποι λέγουν ότι αν είχαν κλείσει τα σύνορα και ήταν αδιαπέραστα, ο πόλεμος θα είχε ήδη τελειώσει. Κύριε Πρόεδρε, εσείς μιλήσατε για προκλήσεις και για εκκλήσεις και για το τι περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι θα πρέπει να ασχολείται ε, και με το θέμα των αστυνομικών δυνάμεων. Εγώ πιστεύω ότι μαζί με εσά και συμφωνώ, δεν φτάνουν πια τα λόγια, έχει φτάσει ο καιρός για τα έργα. Και επιτρέψτε ε, μου να απευθυνθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα προς την κυρία Μόγκερίνη που καμιά φορά έρχεται και να μας δει εδώ ε, και να αρχίσει επιγόντως να ασχολείται με αυτό το θέμα. Φτάνουν τα λόγια. Η Ουκρανία πλέον χρειάζεται έργα. Σλάβα Ουκρανία. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ε, ο συνάδελφος Μαμίκινς. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι έχω μια ερώτηση προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, η ΕΣΤ, η Ουκρανία ήταν η τρίτη μεγαλύτερη ε, πυρηνική δύναμη στον κόσμο. Και όταν ε, το 1994 ήρθε η διακήρυξη της Βουδαπέστης που έλεγε ότι θα είναι ε, αποπυρηνικοποιημένη η Ουκρανία. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση σήμερα αν είχε πυρηνικά η Ουκρανία. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Φωτίγκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εξαιτήμα μέλη της Βερκόφνα Ράντα. Θα ήθελα να επαναλάβω όσα είπα στις αρχές του περασμένου έτους κατά τη συνεδρίαση της ε, κοινής ε, Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ και τη Βερχόπνα Ράντα στο Κίεβο. Δεν έχω καμία αμφιβολία πως ε, τόσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και όσα συνέβησαν στο Μαϊντάν ήταν μια δράση του έθνους που ήθελε να ξεφορτωθεί τους σοβιετικούς περιορισμούς, ήθελε να απελευθερωθεί από αυτή τη ζώνη επιρροής οι νέοι μα έδειξαν ότι με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να περισπίσουν τη χώρα τους. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και οι Ουκρανοί αγωνίζονταν για έναν αγώνα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εμά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Όμως τώρα όλε οι δράσεις που έχουν ε, αναλυφθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία αλλά και από τους ε, αντάρτες ε, ουσιαστικά συνίσταται σε επίθεση στο έδαφος μιας κυρίαρχης χώρας. Αυτό μας αφορά όλους, γιατί πρόκειται για μια απειλή εναντίον όλων μας. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ποιες δράσεις θα αναλάβουμε προκειμένου η Ουκρανία να μπορεί να υπερασπίσει αποτελεσματικά την επικρατειά της. Κύριε Πρόεδρε, στα μέσα του επόμενου μήνα θα στείλουμε μια αντιπροσωπεία στο Κιεβό από την Επιτροπή Σέντε. Εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Αξιολογούμε την κατάσταση ασφάλειας στην Ουκρανία και τις ε, ανάγκες της χώρας. Παρακαλώ να έχετε στο νου σας ε, ότι έχετε 1,5 λεπτό στη διάστησή σας ο κύριος Σε Ευχαριστώ, Αντρέη Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώ ήρθατε σε αυτή την ιστορική επίσκεψη στι Βρυξέλλε του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Είστε φίλοι μα και τέροι μα ε, και σα καλωσορίζουμε. Πρέπει να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθάρρυνε και προώθησε την Ουκρανία να αναλάβει πολλέ μεταρρυθμίσει και να ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή Οδό. Τώρα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να σας βοηθήσουμε σε κάθε περίπτωση. Κύριε Μιλίτα, ε, οι Ρώσοι προσπαθούν να παρουσιάσουν τα γεγονότα στην Ουκρανία, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ουκρανία, σαν έναν εμφύλιο πόλεμο, σαν ε, οι Ουκρανοί να πολεμούν μεταξύ τους για διαφορούς λόγους ξέρω, η Ουκρανική κοινωνία είναι σταθερή και ολοκληρωμένη μπορεί να μιλήσει κανείς ελεύθερα τα στο Κίεβο και δεν ε, θα αντιδράσει κανείς άσχημα. Αντιδρούν φυσιολογικά οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση, να σχολιάσετε την κατάσταση ε, της ε, Κοινωνία στην Ουκρανία, κυρίως για τις μειονότητες. Τι συμβαίνει ακριβώς σήμερα, ποια είναι η σχέση με ε, τις μειονότητες των Τατάρων, των Εβραίων, τη Ρωσική μειονότητα και άλλες που έχετε στη χώρα σας, γιατί μερικές φορές αυτή η εικόνα του εμφυλίου ε, ουσιαστικά έχει αντίκτυπο ακόμη και σε αυτό τον οίκο. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρμς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Κρόισμαν και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έρχεστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά και χαίρομαι που μπορώ να παρευρεθώ κι εγώ. Σήμερα έχω τις εξή δύο ερωτήσεις. Αφού και το Σαββατοκύριακο λίγο πριν ήμουνα στο Σλαβιάν και στο Αρτιμόφσκ και είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω η διεισόμαση ε, της κινήσης ε, των Ουκρανών στρατιωτών και πώς εφαρμόστηκε και χείρια. Ο Υπουργός Εξωτερικών σας εχθές ε, μετέβη στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει και στα Ηνωμένα Έθνη και να ζητήσει και ανόκρανους. Θα μπορούσατε να μας πείτε αυτό πώς συζητιέται στην Ουκρανία και για ποιο λόγο καν έχει ε, προκύψει αυτή η πρόταση. Θα μπορούσατε να πείτε και στους συναδέλφους τι κάνει ο ΑΣΕ, η αποστολή εκεί και πώς εργάζεται και για ποιο λόγο δεν μπορεί αυτή η αποστολή, δεν κατάφερε την περασμένη εβδομάδα να παρατηρήσει ε, τι γίνεται εκεί στην ε, διαχωριστική γραμμή. Επόμενη ερώτηση, ανθρωπιστική κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε ε, φορά ε, προβληματίζεται ε, από τα, τις λευκές αυτοκινητοπομπές από τη Ρωσία προς την Ουκρανία. Τι γίνεται εκεί, πώς το βλέπετε εσείς και τι δράσεις αναλαμβάνετε οι ίδιοι. Ευχαριστώ. Ο εισηγητή μα για την Ουκρανία, κύριος Άριος Βόσκη. Παρακαλώ προσπαθήστε, τσακ να είστε σύντομος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε λίγο θα εγκρίνει την πρόταση μακροοικονομικής βοήθειας 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ε, με ταχεία διαδικασία προς την Ουκρανία χωρίς τροπολογίες και θα διατρανώσει και πάλι την πάγια θέση και δέσμευση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή σε εγκριθεί αυτή η μακροοικονομική βοήθεια θα συνεισφέρει στην υποστήριξη της νόμιμης κυβέρνησης ε, και της Βουλής της Ουκρανίας. Ε, ε, η Βουλή υπό τη δική σας ηγεσία, η κυβέρνηση Ιατσένιουκ και ο πρόεδρος Ποροσέγκο. Για να ε, ελαφρυνθούν κάπως τα οικονομικά που απειλούν ε, την οικονομική σταθερότητα της Ουκρανίας. Δεν είναι φτωχή χώρα η Ουκρανία, αλλά έχει αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση γιατί δεν έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν εδώ και καιρό. Υπάρχει κακή διακυβέρνηση και απώλειες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές λόγω του πολέμου, της ρωσικής εισβολής και κατοχής στη συνέχεια. Χρειάζεται επιγόντως ε, αύξηση και έγκυρη υποστήριξη η Ουκρανία γιατί έχει να αντιμετωπίσει στα ανατολικά την ρωσική εισβολή, ταυτόχρονα αγωνίζεται και παλεύει να σταθεροποιήσει τη χώρα και είναι πρωτοφανέ στην ευρωπαϊκή ιστορία μια, Ευρώπη, μια χώρα στην Ευρώπη που έχει τέτοιε τεράστιε προκλήσεις να αντιμετωπίσει, τι αντιμετωπίζει ταυτόχρονα. Είναι και αποσταθεροποιητική η κρίση και οικονομικά και χρηματοοικονομικά και εν μέρος αυτό οφείλεται ε, γιατί ε, ε, είναι όμοιρος μέχρι και το 20% της οικονομίας για την άμυνα της χώρας. Το καλύτερο δώρο που έχει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνή κοινότητα προς τον εισβολέα, τη Ρωσία και τον ίδιο το Πούτιν θα ήταν να επιτρέψει την πτώχευση τη χροκοπία της Ουκρανίας, πράγμα που δεν πρόκειται εμείς να επιτρέψουμε. Κοιτάξτε, οι υπόλοιποι πέντε συνάδελφοι να Είστε σύντομοι, γιατί στι 4 ο πρόεδρο Γκρόσμαν θα πρέπει να πάει να δει τον κύριο Σούλτ. Ένα λεπτό το πολύ έκαστος, τουλάχιστον για να απαντήσει ο πρόεδρο. Ο κύριο Μπαλτσίτης, παρακαλώ. <clears throat> Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ακούσαμε ήδη πολλέ ιδέε και εσεί, κύριε πρόεδρε και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει είναι εκτό πραγματικότητα. Εγώ εκπροσωπώ τη Λιθουανία Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι από άλλες χώρες της Βαλτικής και όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε τι εστί σοβιετική κατοχή και τι χρειάζεται μετά, τι χρειάστηκε για να αναπτυχθούν οι οικονομίες μας. Εμείς όλοι υποστηρίξαμε την Ουκρανία, όπως γνωρίζετε. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική σήμερα στην Ουκρανία. Δεν μπορούσαμε να την είχαμε φανταστεί ούτε κατά διάνοια πριν από λίγα χρόνια ήταν πολύ ψηλή και η διαφθορά στη χώρα και μετά από δεκαετίες ε, τέτοιων καταστάσεων ε, έχει αφήσει πολύ άσχημη κληρονομιά. Τώρα ακούσαμε για την χρηματοοικονομική βοήθεια που θα δοθεί, μάλλον συμβολικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση ε, επαρκής. Θα ήθελα λοιπόν κύριε Πρόεδρε της Ράντα να σας ρωτήσω πόσο καιρό θα μπορέσετε να επιβιώσετε με τέτοιο είδους συμβολική υποστήριξη της Δύσης και απουσία της παράδοσης όπλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να υποστηρίξω τον κύριο Παροσένκο, ο οποίος ε, κάνει έκκληση να υπάρξουν διεθνείς συνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Το έχω πει και στο παρελθόν και θα το ξαναπώ. Πρέπει να απαντήσουμε θετικά σε αυτό το αίτημα. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξει αυτή την πρωτοβουλία. Το συντομότερο αυτό είναι ο ρόλο και το καθήκον μα και είναι και εντό τη δικαιοδοσία μα. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Ποια ήταν ε, η απάντηση από την Ουκρανική κοινωνία και από τα μέλη της κυβέρνησης σε αυτό το αίτημα του κ. Ποροσένκου και πώς αντίδρασαν και τα κοινοβούλια στο εξωτερικό. Και μια άλλη ερώτηση. Ο Δησός και το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, ε, η ακτή της Μαύρης Θάλασσας, εκεί σε αυτές τις περιοχές είναι ασφαλής η κατάσταση ή μπορεί να υπάρξουν και εκεί κάποιες απειλές. Και τώρα, κατόπιν τόσο ακούσαμε και από τους προηγούμενους ομιλητές για τους ε, τάρους της ε, Κρυμαίας. Ε, Υποστηρίζεται τα δικαιώματά τους παρόλο που βρίσκονται υποκατοχή. Ευχαριστώ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου υπόθηκε ότι η Ομοσπονδίση θα οδηγήσει την Ουκρανία σε κατάρρευση ενώ συγκεντρωτισμός επιτυχία με τη συμφωνία των 12 σημείων ε, και ενώ καλείται η Βουλή σε 30 μέρες να δώσει στις περιοχές του Λουμπάκ και του Ντονέσκ μια εντολή αυτοδιακυβέρνησης, στο πλαίσιο αυτό βλέπετε αυτή την προσωρινή εντολή ως μια πολιτική ανοιχτή πόρτας ε, προκειμένου οι περιοχές των αυτονομιστών να κηρύξουν την ε, αυτονομία και εν τέλει ε, θα οδηγηθούμε σε ομοσπονδιοποίηση της Ουκρανίας ή σε ένα δημοψήφισμα για ανεξαρτησία και μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει με τις μελλοντικέ εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2015. Παρ' όλα αυτά, αναμένεται μια δυνατότητα μποϊκοταρίσματος των γενικών εκλογών ή μια αναγνώριση των αποτελεσμάτων στο Ντομπάς και στο Λουγκάνσκ όπου εκεί μπορεί να γίνουν εκλογές από τους ρωσόφιλους, ο κ. Παπαδάκης. Κύριε Γκρούσμαν, στη χώρα σας ο κ. Μπρόγκ ε, είπε ότι τίνει να γίνει υπόδειγμα προς μίμηση η χώρα σας. Με προκλητικό τρόπο η κυβέρνηση που στηρίζεται και από φασιστικές δυνάμεις πολιτικά διέλυσε την κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας. Παράλληλα παρετήθηκε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου του Κιέβου γιατί υποβλήθηκε σε έρευνα στα γραφεία του σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε άλλα προσωπικά του αντικείμενα. Αυτά, αυτές οι έρευνες έγιναν και σε άλλους ε, δικαστές. Άλλοι δέκα δικαστές μάλιστα ζήτησαν εξαίρεση από την δίκη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας. Και λέμε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που επικαλείται υποκριτικά και επιλεκτικά τα δημοκρατικά δικαιώματα, όποτε θέλει τα χρησιμοποιεί σαν πρόσχημα για εμπεριληστικές επεμβάσεις όπως έγινε στην Ουκρανία, για συμφέροντα των μονοπωλίων και έχει και υπογράψει και συμφωνία σύνδεση με την αντιδραστική Ουκρανική κυβέρνηση. Πώ τοποθετήσετε, κύριε Γκρούσμαν, στην δίωξη του Κομμουνιστικού Κόμματο Ουκρανία, στη διάλυση τη κοινοβουλευτική του ομάδα και στι προκλητικέ μεθοδεύσει στη δίκη παροδία που γίνεται σε βάρο του Κομμουνιστικού Κόμματο Ουκρανία, πρέπει να απολογηθείτε. Thank you. Uh, and the final speaker is Mr. Nart. Νάρτ, Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι... Ορίστε. Ε, η σειρά μου δεν είναι μάλιστα. Έλεγα, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου φίλο της Ουκρανίας και είμαι και στην ομάδα φιλίας της Ουκρανίας. Αλλά στους φίλους θα πρέπει να λέμε ειλικρινά τι πιστεύουμε και όχι απλώς να μην διούμε. Έχω μερικές ερωτήσεις που με ε, προβληματίζουν. Η Ουκρανική πατρίδα κινδυνεύει και υπήρξε εισβολή στην Κρυμαία και αρχίζει να αποσχίζεται στο Ντονέσκ. Στις εκλογές πηγαίνουν να ψηφίσουν μόνο οι μισοί Ουκρανοί, δηλαδή 52%. Οι υπόλοιποι μένουν σπίτι τους. Έχω εδώ δηλώσεις ε, του Υπουργού Αμήνης της Ουκρανίας που είναι ε, αντιστράτηγος ε, και λέγει ότι μόνο το 20% των στρατιωτών θέλησαν να πάνε στο μέτωπο που υπηρετούσαν τη θητεία του σε καιρό πολέμου. Δεύτερη ερώτηση. Θεωρεί, μάλλον το 1991 αποκτά την ανεξαρτησία της η Ουκρανία. Πώς είναι δυνατόν να χρειάζονται πολιτοφυλακές που να τις πληρώνουν ολιγάρκες όπως είναι και στο Ντονέσκ και στο Λουχάνσκ. Ε, δεν είναι διαφορετική η κατάσταση. Τρίτο ερώτημα που με απασχολεί. Εγώ είμαι δημοκράτης. Ε, το, η πολιτική ε, δεν ε, ταυτίζεται με τις business. Πώς γίνεται οι οικονομικοί ολιγάρχες να είναι και πολιτικοί ηγέτες από τον Ποροσέγκο αρχής γενομένης μέχρι τον Κορομόσκι και από την άλλη ο Πακολίν και ο Κοημόν. Πώς είναι δυνατόν να είσαι ολιγάρχης και να λες ότι θες να πατάξεις τη διαφθορά. Ναι, ευχαριστώ. Νομίζω καταλάβαμε τι θέλετε να πείτε. Έχετε το λόγο κύριε Γκρόσμα για να συνοψίσετε. Παρακαλώ. 5-6 λεπτά. Ε, Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ειλικρινή συζήτηση, για τις ειλικρινείς ερωτήσεις και για τις θέσεις που υιοθετείτε, γιατί αυτές είναι σημαντικές για την Ουκρανία. Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι υφιστάμεθα μία επίθεση άνευ προηγουμένου όχι μόνο στο στρατιωτικό σκέλος αλλά και στο οικονομικό σκέλος και στο σκέλος της πληροφόρησης αλλά και της ενέργειας. Δυστυχώς αυτό στρεβλώνει και τις εξελίξεις τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία. Δεν είναι μυστικό το ότι σήμερα στην Ουκρανία οι ειδικέ δυνάμεις που έχουν εκπαιδευτεί και προετοιμαστεί από τις ειδικέ δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν πολύ βαρύ οπλισμό που προέρχεται από τη Ρωσία. Δεν υπήρχε λόγος για εσωτερική σύγκρουση στην Ουκρανία. Μιλήσατε για την ομοσπονδιοποίηση. Γιατί να χωρίσουμε μια χώρα η οποία ήταν ενωμένα, ενωμένη. Μιλάτε για αυτονομία. Φίλοι μου, θυμηθείτε ότι η κατεχόμενη Κρυμαία ήταν αυτόνομη δημοκρατία της Ουκρανίας. Παρόλα αυτά, δεν σταμάτησε ο, ο επιτιθέμενος. Φαίνεται ότι κάποιος κάτι μπορεί να θέλει από μας και εμείς έχουμε την πραγματική μας βούληση. Και ποια είναι η βούλησή μας. Εν πάση περιπτώσει οι δημοκρατικές αξίες, η δαφική ακεραιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε στην αρχή αξιολογώντας την κατάσταση ότι πρέπει να αποκαλέσουμε τα πράγματα με το όνομά τους και συμφωνώ απολύτως για να μπορέσουμε τελικά να δράσουμε. Είμαστε ανοιχτοί, θέλουμε ειρήνη και θέλω να τονίσω ότι είμαστε και έτοιμοι για ειρηνική επίλυση. Δεν θέλουμε πόλεμο. Εμείς δεν επιτεθήκαμε σε κανέναν. Και δεν θα επιτεθούμε και σε κανέναν στο μέλλον. Θέλουμε η Ουκρανία να είναι κυρίαρχη χώρα. Δεν θέλουμε ο πληθυσμός, ο άμαχος πληθυσμός να πεθαίνει, ούτε οι στρατιώτες μας. Αυτό είναι πρόκληση. Ο επιτιθέμενος δεν θέλει μόνο την Ουκρανία, θέλει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να πιστέψουν ότι αυτά τα οποία πιστεύουμε εμείς δεν σημαίνουν τίποτα. Θέλει να δείξει σε όλη την Ευρώπη ότι το δίκαιο είναι με το μέρος του ισχυρού. Ο επιτιθέμενος όμως Πούτιν θα σταματηθεί. Το ερώτημα είναι πότε. Τώρα, ω προ και την τωρινή μα αντίδραση, ο Πρόεδρο, ναι, ανέλαβε την πρωτοβουλία για Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλεια και ζήτησε αποστολή για τη διατήρηση τη ειρήνη. Και η αποστολή αυτή θα μα επιτρέψει να σταματήσουμε τι επιθέσει και μα είπαν ότι πρέπει αυτό να είναι στη γραμμή του μετόπου αλλά και στα σύνορα. Πρέπει να είναι παρόντες ή της αποστολής διατηρήσης της ειρήνης. Και βεβαίως υπάρχουν κυρώσει. Και δεν πρέπει να τιμωρούμε την πίεση. Η πίεση είναι η διαντίδρασή μας για να σταματήσουμε την επίθεση που υφιστάμεθα. Εγώ ενδεχομένως είμαι αυτός που λιγότερο από όλους θέλει τις πιέσεις, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει να ασκήσουμε αυτή τη πίεση. Και ένα άλλο σημαντικό είναι ε, οι αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας. Πότε μόνο όταν θα πάρουμε ε, τα, τον οπλισμό τον αμυντικό που είναι επαρκής, μόνο τότε θα σταματήσουμε τον εχθρό ο οποίος προχώρησε στο ουκρανικό έδαφος και θέλει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο και γι' αυτό η ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας είναι εξαιρετικά ε, ε, σημαντική. Τώρα, έχουμε ξεκινήσει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Οι εσωτερικές μεταρρυθμίσεις για όλες τις ομάδες ε, τις είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Και με αυτό το στόχο έχουμε εκλεγεί, εκλεγεί να αλλάξουμε τη μετασοβιετική Ουκρανία, ούτως ώστε να γίνει μια αληθινά ευρωπαϊκή χώρα, να σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων ε, των ε, πληθυσμών, να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, να έχουμε ε, σωστή δίκαιη δικαιοσύνη. Και θα το κάνουμε. Χρειαζόμαστε χρόνο, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Αυτό το παράθυρο ευκαιρίας είναι ανοιχτό για σύντομο χρονικό διάστημα. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν αναθεώρησης του συντάγματος θα δουλέψουμε πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα, ως προς το σχέδιο ειρήνευσης, αυτό προτάθηκε και περιλαμβάνει τα πάντα, την κατάπαυση του πυρός, την απόσυρση του βαρέως οπλισμού από τα μέρη, την απελευθέρωση όλων των ε, κρατουμένων ε, στρατιωτών που βρίσκονται στις φυλακές της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων, των οποίων βρίσκεται και η κυρία Σαπτσέγκο. Και μετά από τις τοπικές εκλογές του 2010, στο Ντόνετσκ και αλλού, η κυβέρνηση η οποία είχε νομίμως εκλεγεί εξαναγκάστηκε να φύγει. Το δημοψήφισμα είχε γίνει με τη βοήθεια των όπλων. Δεν ανταποκρίνεται στη βούληση του κόσμου που ζει εκεί και υποφέρει. Ουσιαστικά κρατείται ο κόσμος παρά τη θέλησή του εκεί. Κοινός μας στόχος είναι να πολεμήσουμε τον εχθρό, να δώσουμε αυτό τον αγώνα υπέρ των ευρωπαϊκών αξιών, να κάνουμε τα πάντα για να έχει ειρήνη η χώρα μας όχι μόνο στα χαρτιά αλλά και στην πραγματικότητα. Η πραγματική ειρήνη, η αληθινή ειρήνη, αυτή είναι η εγγύηση Ξέρετε, πάρα πολλές ερωτήσεις μου έχουν τεθεί, δεν έχω χρόνο να τις απαντήσω όλες. Ως προς τις ε, ε, εθνοτικές μειονότητες μπορώ να σας πω το εξής. Καταθέτω ότι η Ουκρανία δίνει αγώνα υπέρ των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Η Ουκρανία είναι μια χώρα με πολύ μεγάλη ανεκτικότητα Έχουμε όμως και τσετσένους μαχητές οι οποίοι δεν είναι Ουκρανοί, οι οποίοι είναι εχθροί. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μου των συναδέλφων από την Ουκρανία για την προσοχή που δίνετε στο ουκρανικό θέμα για την πολύ σημαντική θέση που υιοθετείτε και την οποία στηρίζουμε σήμερα. Ζήτω η Ουκρανία σε μια ε, δημοκρατική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you very much, President Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρόισμαν. Καταφέρατε να απαντήσετε τα περισσότερα ζητήματα. Νομίζω ε, όλοι χαρήκαμε για την ευκαιρία που είχαμε να αλλάξουμε απόψεις μαζί σας. Και τώρα οι υποχρεώσεις σας σας ε, καλούν στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, θα τα πούμε στη συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Δεν είπατε τίποτα για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν είπατε τίποτα σας έκανα ερώτηση και δεν απαντήσατε. Σε ό,τι αφορά για τα κόμματα, σε ό,τι αφορά στα κόμματα, θα ήθελα να σας πω για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εμείς θα πρέπει να στήσουμε ένα δημοκρατικό σύστημα με διαφάνεια, με εμπιστοσύνη σε όλα τα κόμματα. Αλλά θα ήθελα να πω ότι για πρώτη φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα έμεινε εκτός Κοινοβουλίου και αυτό λέει πολλά για την ευρωπαϊκή επιλογή μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Let us continue with the... Ε, συνεχίσουμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξή μας τώρα. Είμαστε στο σημείο 17 για την μακροοικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σας ζητήσω λίγη ησυχία, κοιτάξτε. Like to leave uh, the room, please do it so in quiet. Όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, παρακαλώ το πράξτε εισήγως. Είναι πολύ φορτωμένη η ημερήσια διάταξή μας και πρέπει να συνεχίσουμε. Άρα λοιπόν, είναι γνωμοδότηση προ την ΙΝΤΑ για τη μακροοικονομική συνδρομή στην Ουκρανία. Συντάκτη γνωμοδότησης είναι ο κύριο Σάριο Βόλσκι. Η Ουκρανία, όπω γνωρίζουμε και ακούσαμε στη συνεδρία και στη συζήτηση, χρειάζεται ακόμα τη βοήθειά μα για να αντιμετωπίσει την τόσο μεγάλη κρίση που έχει και την οικονομική. Και επειδή μειώνονται σε οξύτατο βαθμό οι ξένε επενδύσει. Προτείνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1,8 δις επιπλέον μακροοικονομικής βοήθειας, ε, ε, ε, επιπλέον του πρώτου δανείου του 2014 που ήταν 1,6 δις. Η τελευταία δόση θα καταβληθεί το Μάρτιο. Η Λετωνική Προεδρία έχει ενημερώσει την επί της αρμόδια επιτροπή ότι δεδομένης της επίγουσας κατάστασης στην Ουκρανία έχει συμφωνήσει ε, το Συμβούλιο βάσει των αρχικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς τροπολογίες. Και το ίδιο ε, θα γίνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Σάριος Βόλσκι για να εξηγήσει λεπτομέρειες την πρότασή του αυτή και πάλι. Προτείνω uh, η Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων να, να υποστηρίξει ένθερμα αυτή την ε, ταχεία διαδικασία γιατί οι ανάγκες της Ουκρανίας ε, είναι άμεσες. Επομένως, αυτή η ταχεία διαδικασία χωρίς τροπολογίες ε, θα είναι μια επιβεβαίωση δεσμευσή μας να λάβει η Ουκρανία το ποσό που αναφέρεται. Μιλάμε για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων σε μια κατάσταση όταν ε, η ε, κακή οικονομική κατάσταση χώρας ε, έχει επέλθει όχι μόνο λόγω της προηγούμενης κακής διαχείρισης της, της προηγούμενης κυβέρνησης αλλά και λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Επομένως, πλήρη υποστήριξη της Επιτροπής μας θα πρότεινα σε αυτή την επιταχυνόμενη διαδικασία και την απόφαση να δώσουμε αυτή τη μακροοικονομική βοήθεια στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, κατά την άποψή μου, τονίζω στην γνωμοδότησή μου ότι είναι απαραίτητη αυτή η βοήθεια να είναι όσο και να είναι όσο το δυνατόν πιο γενναιόδορη και να προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει και άλλους τρόπους να διευκολύνει την οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας και τα κράτη-μέλη να τη διευκολύνουν με διάφορα διοικητικά μέσα και προκειμένου να επιστραφούν στην Ουκρανία όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία παράνομα κατήχε ο Γιαννούκοβιτς και τα οποία τώρα είναι κρυμμένα στις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν μπορούσε να ανακτήσει η Ουκρανία αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, αυτά να μην ε, σταλούν για να ικανοποιήσουν ε, αξιώσεις των Ρώσων, αλλά να καλύψουν τις ανάγκες του κρανικού κράτους. Επίσης προτείνω θα πρέπει να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ε, προσπάθεια της Ουκρανίας να καταπολεμήσει την ενδυμική διαφθορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει ένα κοινό ερευνητικό όργανο που θα παρακολουθεί την χρηματοοικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία. Αυτός ο φορέος όχι μόνο θα διασφάλιζε ότι θα δαπανόνταν σωστά τα κονδύλια, αλλά και ότι ε, θα χρησιμοποιούνταν για το να ε, υπάρχει οικοδόμηση θεσμών ε, και να υπάρχει και οικονομικός έλεγχος και λογιστικός έλεγχος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να στηρίξει τα πιο ευάλωτα τμήματα της ουκρανικής οικονομίας, ενέργεια, επιχειρησιακό περιβάλλον, φορολογία και φορολογική πολιτική και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεισφέρει στο να αμβλύνει τις δυσκολίες της Ουκρανίας. Και μπορώ να πω ότι ένας φίλος την ανάγκη φαίνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να είναι ένας φίλος προς την Ουκρανία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Γιάτσεκ. Είναι καλό ότι και αρκετοί συνάδελφοι από τη Βέρχον Ράντα ήταν εδώ, όταν εξήγησα σε αυτή τη θέση. Δεν βλέπω να ζητούν συνάδελφοι το λόγο. Έτσι λοιπόν, αυτό σημαίνει όπως ε, και στο Συμβούλιο σημαίνει ότι και οι βουλευτές εδώ έχουν καταλάβει ότι εδώ πρόκειται για μια ταχεία διαδικασία, χωρίς τροπολογίες και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι όλοι υποστηρίζουμε ένθερμα αυτό το νέο σκέλος οικονομική συνδρομή στην Ουκρανία. Ένα σύντομο σχόλιο από την Κομισιόν. Ο κ. Γιάννη Γκρίσεν είναι εδώ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά η Κομισιόν καλωσορίζει την υποστήριξη που εκφράζεται από την Επιτροπή σας, όπως ε, και από χθε, από την Επιτροπή ΙΝΤΑ, την Καθήλια Αρμοδία Επιτροπή και απλώς θέλω να τονίσω το κατεπήγον του φακέλου αυτού. Η Ουκρανία βιώνει μία μακρά και βαθιά ύφηση. Ε, έτσι λοιπόν ακριβώς ε, Γι' αυτό η πρότασή μας μικροοικονομικής συνδρομής ενός ακόμη πακέτου, μιας ακόμη δεσμής μέτρων, έχει ως στόχο να ανακουφίσει αυτή την πολύ σοβαρή κατάσταση. Είναι μέρος ενός ευρύτερου διεθνούς πακέτου για την Ουκρανία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προετοιμάζει ένα πακέτο αρρωγή 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων όπου έχουμε συνεισφορές από το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διμερείς συνεισφορές όπως η δική μας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ιδιωτικό τομέα, μπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Έτσι λοιπόν έχει ανακοινώσει η Ουκρανική κυβέρνηση ότι θα αρχίσει διαβουλεύσεις ε, ε, με τους πιστωτές της ε, για να μπορεί να παρατείνει την διάρκεια αυτών των χρεών και επίσης να δούμε και πώς θα διασφαλιστεί η χρηματοδότηση της χώρας τα επόμενα έτη. Θα περιοριστώ σε αυτά, καλωσορίζουμε την υποστήριξή σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκρίσε. Να επενθυμίσω σε όλους τους συναδέλφους τουλάχιστον επίσημα, ότι έχουμε μια προθεσμία κατά τροπολογίων 26 Φεβρουαρίου, αλλά όπω είπαμε δεν θα έχουμε τροπολογίε. Έτσι λοιπόν εδώ ολοκληρώνουμε το σημείο 17 τη ημερησία διάταξη και θέλω να ζητήσω στο, από τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Πάσκο, να αναλάβει την Προεδρία. Πάμε μέσα στο επόμενο θέμα. Ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων Κασιτέρου, Τανταλίου και Βολφραμίου, των μεταλλαγμάτων τους κτλ. Εισηγητής είναι εδώ ο κύριος Κόφερ, συντάκτης γνωμοδότης για την ακρίβεια, ο οποίος έχει το λόγο αμέσως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων αυτή. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που με κατέκλυσαν με τροπολογίες. Προσκαλώ τους και τους στη συνεδρίαση στις 26 Φεβρουαρίου και ελπίζω να μπορέσουμε να τα βρούμε. Διαδικαστικά μέχρι στιγμής μία είναι η δυνατότητα στον προγραμματισμό προβλέπεται να ψηφιστεί το σχέδιο της νομοδότησης εδώ στην Επιτροπή μας στις 9 Μαρτίου. Ωστόσο, επειδή η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΙΝΤΑ έχει αναβάλει τη δική της ψηφοφορία στις 13 και 14 Απριλίου είναι πλέον. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να βρούμε και περισσότερες συμβαστικές απολογίες, αν το επιθυμούμε. Αυτό βέβαια θα το αποφασίσει το Προεδρείο, αλλά το θέτω υπόψη σας. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε για δεύτερη φορά στις 9 Μαρτίου, να ψηφίσουμε. Προχωρώ στη γνωμοδότηση τώρα αυτή καθ' αυτή. Όπως σας γνωρίζετε όλοι, είναι υποθέτεται, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ αμφιλεγόμενο. Και αυτό άλλωστε έχει υπογραμμιστεί και από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Ορισμένε είναι πιο χαλαρέ από τις δικέ μου προτάσει. ενώ κάποιες άλλε σε περίπτωση που ευδοκιμήσουν θα είναι πιο ε, αυστηρές, α πούμε, από το σχέδιο της δική μου γνωμοδότησης. Ουσιαστικά εγώ τι προσπάθησα να κάνω. Να μείνω στη μέση οδό ε, τηρώντας ε, την νομοθεσία Dodd-Frank ε, που έδωσε πολλές ιδέες για τη δική μας δουλειά. Μιλώ για την Αμερικανική νομοθεσία. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασιστήκαμε για τη χάραξη της δικής μας πρότασης. Τι σημαίνει αυτό. Just on importers. Ότι δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στους εισαγωγείς και στην εθελούσια συνεργασία. Το σχέδιο γνωμοδότησης ομιλεί για υποχρεωτική δήλωση και αναφορά και περιορίζει το πεδίο εφαρμογή ε, του προτινόμενου κανονισμού. Πάρα πολύ κοντά στην προσέγγιση τύπου Dot Frank. Προφανώς η δική μας επιτροπή θα πρέπει να επιλέξει τη δική της στρατηγική, αλλά Προσωπικά πιστεύω ότι συχνά ε, μιλάμε για κανονιστικές ρυθμίσεις και εναρμόνιση όσο γίνεται περισσότερο στο διατλαντικό ε, πεδίο συνεργασίας. Νομίζω καλό θα ήταν εδώ να ε, προχωρήσουμε περισσότερο προς την εναρμόνιση. Φυσικά μου έκαναν κρούσεις διάφορα λόμπι που έλεγαν ξεκάθαρα ότι ήθελαν ασθενή ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ πιο ασθενή από την Dot Frank, για να τη χρησιμοποιήσουν αργότερα ως μοχλό για να υπονομεύσουν ε, ή για να παρακάψουν τον Dot Frank στις διατλαντικές διαπραγματεύσεις. Και από την άλλη υπάρχουν και κάποιοι άλλοι και οι συνάδελφοι θα πούν τη δική τους γνώμη που ελπίζουν να έχουν πιο ε, υψηλότερο επίπεδο ρυθμίσεων και προτύπων από ότι το συστημα dot Dodd-Frank. Θα δούμε τι θα βγει από όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά ήθελα να το αναφέρω. Και ο φετινός ε, κάτοχος του γραφείου Σαχάροφ, ο δόκτωρ Μοκουέγε, προειδοποίησε το Κοινοβούλιο και είπε ότι θα πρέπει να ε, γίνει η νομοθεσία αυτή υποχρεωτική ανάλογη της νομοθεσίας Dodd Frank των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ποιες είναι οι πολιτικές γραμμές που θα πρέπει να αποφασίσουμε εμείς, χονδρικά. Το είπαμε ήδη, το σύστημα θα είναι θελοντικό ή υποχρεωτικό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση συναδέλφων του ΕΛΚ που λέγει ότι κάπως θέλει τα δύο να τα συνδυάσει. Για την περιοχή των μεγάλων ε, λιμνών να είναι υποχρεωτικό, αλλά για τα υπόλοιπα μέρη να είναι θελοντικό. Και υπάρχει και το θέμα της γεωγραφικής έκτασης και του πεδίου της γεωγραφικής εφαρμογής. Ε, καλό είναι να γνωρίζουμε και είναι θετικό αυτό ότι φαίνεται ότι ε, συμφωνούν όλες οι πλευρές ότι δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε κάποια γεωγραφική περιοχή αλλά να είναι εκτενές. Επίσης, ένα θέμα, αν θα αφορά μόνο τους εισαγωγείς ή γενικότερα τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί. Και επίσης είναι και το θέμα των πόρων, δηλαδή θα πρέπει να μείνουμε σε αυτά τα τέσσερα στοιχεία ε, που συνδέονται με περιοχές που είναι σε σύραξη ε, που στα αγγλικά έχουν αρχικά τα τρία πρώτα ταφ και το τελευταίο G ε, που είναι δηλαδή ταντάλιο, κασίτερος, βολφράμιο και χρυσός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουτικόφερ και τώρα θα παρακαλέσουμε τους επόμενους ομιλητές, ο κ. Αντάξουτσον που είναι και σκιώδης εισηγητής επίσης. Ε, Ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπουτικόφερ ε, για το έργο του. Πρέπει να αναγνωρίζουμε ε, ότι στην Επιτροπή υπάρχει συμφωνία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξοι όταν μιλάμε για την καταπολέμηση των αιτιών αυτής της ε, σύραξης και φυσικά ε, ξέρετε η ύπαρξη αυτών των μεταλλευμάτων ε, κάνει να θεωρείται αυτές τις περιοχές από τις πλουσιότερες αλλά εν τέλει είναι μία από τις φτωχότερες και ότι βγαίνει από εκεί πηγαίνει ε, στην πιο πραγματική τεχνολογία, στα κινητά τηλέφωνα, στους υπολογιστές κτλ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν ότι υπάρχει δίκαιο ηθικό εμπόριο αυτών των μεταλλευμάτων αλλά και των προϊόντων που τα περιέχουν πρέπει να υπάρχει ανιχνευσιμότητα και διαφάνεια. Αυτές πρέπει να είναι κατευθυντηρίες γραμμές. Οι συνέπειες ενός ε, νέου συνόλου κανόν εργορίου για αυτά τα μεταλλεύματα δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι μιλάμε για παγόρευση, μποϊκοτάζ αυτών των μεταλλευμάτων. Αυτό θα έπλητε τους ντόπιου πληθυσμούς. Αντίθετα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα βάλουμε ένα τέλος στην παράνομη εξόριξη που ε, καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση των ένοπλων ομάδων. Εδώ, ε, αν ε, θέλουμε να προωθήσουμε την νόμιμη εξόριξη την μεταλλευτική δραστηριότητα ε, με ε, αξιοπρεπείς μισθούς θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και τα έσοδα του μεταλλεύματα φτάνουν στον τοπιο πληθυσμό. Θα πρέπει να πιέσουμε για νομοθεσία που συνεισφέρει στη διαφάνεια και για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και για τους καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα θα δίνει και κίνητρα να υλοποιηθεί αυτό το ηθικό εμπόριο που θα ωφελήσει τους ντόπιου πληθυσμού. Αυτό θα είναι κινήτρο να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει πλέον βία στις σειράξεις και το εγώ σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες προς αυτό το πνεύμα. Καταρχήν, Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη συνεργασίας ε, μεταξύ ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΟΣΑ και Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να έχουμε ένα παγκόσμιο καθεστώς και θέλουμε και υπεύθυνα μεταλλουργία και καταστάσεις εξευγενισμού που να καλύπτουν το 80% του συνόλου προκειμένου να δώσουμε και στις εταιρείες κατάντη στην αλυσίδα μια βεβαιότητα σε σχέση με τα μέτρα που θα ισχύουν και ότι θα μπορούν να συνεχίσουν την εμπορία ε, μεταλλευμάτων από την ε, ε, περιοχή των Μεγαλών Λιμνών και το Κονγκό. Δεν έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή ένα κατάλογο των υπεύθυνων μεταλλουργίων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού, αλλά αυτό θα σήμαινε ότι θα είχαμε μειονεκτήματα για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε χωρί να βελτιωθεί η κατάσταση στην αγορά. Δεύτερον, οι λόγοι για αυτό το εθελούσιο σύστημα θα πρέπει παρόλα αυτά να είναι υποχρεωτικό για του εισαγωγεί των μεταλλευμάτων που καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού και μιλάμε για τα μεταλλεία που έρχονται από την περιοχή των Γαλλιμνών και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Αυτή η πρόταση προσπαθεί να βασιστεί στο η δουλειά που είχε ξεκινήσει βάσει της νομοθεσιας Dot Dodd-Frank και επίσης προσπαθεί να διαχωρίσει τα καθαρά τα μεταλλεύματα που έρχονται από όλες περιοχές από τα μεταλλεύματα που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες. Πρέπει να υπάρχει βελτίωση εντός της αλυσίδιας εφοδιασμού και Επίσης πρέπει να μπορεί κάποιο να αγοράζει μεταλλεύματα και να ξέρει ότι δεν χρηματοδοτεί πλέον τι σειράξει. Ευχαριστώ κύριο Να. Ευχαριστώ. Για μένα ο πολεμός δεν είναι απλώς μια αναφορά που διαβάζω στις εφημερίδες ή βλέπω στην τηλεόραση. Για 25 χρόνια ήμουν πολεμικός ανταποκριτής και από την εμπειρία μου ξέρω ποια είναι η βαρβαρότητα και από πού πηγάζουν οι πόλεμοι και η χρηματοδότηση. Εγώ έχω υποβάλει διάφορες τροπολογίες ε, στο σχέδιο με την ακόλουθη μορφή. Ε, διακίνηση των φυσικών πόρων είναι ο λόγος για την τρομοκρατία, για τα παιδιά στρατιώτες, για τη σκλαβιά ε, στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι ε, οι κοινωνίες που θέλουν να πλουτίσουν θα αυτορυθμιστούν και χρειάζεται μια αυστηρή ρύθμιση που να εμποδίσει να συνεχίζεται αυτή η τρομερή ρεγοδία στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και που ε, καταλήγουμε στο να είναι συνένοχες και χώρες και εταιρείε που έχουν ε, θέσει σε εμπορία αυτά τα μεταλλεύματα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την υποκριτική στάση ότι θα, ε, θα κλείνουμε τα μάτια μας στην προέλευση στρατηγικών μεταλλευμάτων για λόγους εμπορίου. Και δεύτερο, ένα, δεύτερο, ένα άλλο σημείο που πρέπει να σκεφτούμε είναι τα τελικά προϊόντα που υλοποιούνται κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες. Η Κίνα, παραδείγματο χάρη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαιτήσουμε οποιοδήποτε προϊόν που έχει κατασκευαστεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός από το διάβλο ελέγχου και εισαγωγή, αλλά και θέση σε εμπορία ή των ίδιων των μεταλλίων να έχει ένα πιστοποιητικό καθαρή προέλευση. Διαφορετικά να μην επιτρέπουμε την εισαγωγή. Αυτό για διτό λόγο. Για να μην επιτρέψουμε να συνεχιστεί σφαγή και θάνατη που γίνονται από τις άλλες χώρες ε, και επειδή οι δικοί μας μηχανίες δεν θέλουμε να ζημιωθούν από τον ανταγωνισμό, από τα πιο φτηνά μεταλλεύματα που θα έχουν αποκτηθεί με εγκληματικό τρόπο. Εγώ ειλικρινά την πρόταση της Κομισιόν που ζητά την εκούσια αυτορύθμιση τη θεωρώ υποκριτική ουτοπική. Είναι σαν να ζητούσαμε ε, ουσιαστικά από... Ε, από το μαστροπό να αυτορυθμίσει ε, την πορνεία, την εμπορία ανθρώπων. Ουσιαστικά φαίνεται σαν να αφήνουμε μια δυνατότητα διαφωγή, σαν αυτοί που μπορούσαν να ξεφύγουν από την νομοθεσία Dot Frank των ΗΠΑ να, μπουν, να βάλουν τα μεταλλεύματα αυτά δια της Ευρωπαϊκής Οδού. Όμως το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν μπορούμε να δεχτούμε την αυτορύθμιση γιατί είναι η οδός προς την απάτη και δεν αξίζει τότε να ζητήσουμε τίποτα. α πούμε ότι δεν μα ενδιαφέρει, ασφαγιάζονται οι λαοί στους τόπους προέλευση, ε, αν το εμπόριο πάει καλά. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πολύ, ο Στάνοκ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μπιούτι Κόφερ για τη σημαντική δουλειά που έχει κάνει, γιατί το θέμα είναι δύσκολο, ακαθόδης και αμφιλεγόμενο και έχει και πολλά συμφέροντα εδώ. Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα χρόνια την επιτυχία της διαδικασίας Κίμπερλι, τα διαμάντια ε, βουτυγμένα στο αίμα από τη Δυτική Αφρική. Και έχει ενδιαφέρον που ε, αυτό επεκτείνεται και σε άλλα μεταλλεύματα από περιοχές σε σύραξη. Και στην Αφρική ε, βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο τα διαμάντρια και άλλες πλούτοπαραγωγικές πηγές έχουν ε, ε, χρηματοδοτήσει τις πιο αιμοσταγείς πολιτοφυλακές. Ταντάλιο, χαλκός και τα λοιπά δεν είναι μόνο αυτά που αναφέρονται εδώ. Χαίρομαι λοιπόν ε, για την πρόταση αυτή. Το θέμα είναι αν θα πρέπει να είναι τώρα εθελοντική, αυτή η αυτορύθμιση, αυτοπιστοποίηση ή υποχρεωτική. Οι Αμερικανοί ε, έχουν μέχρι τώρα την πιο αυστηρή νομοθεσία ε, δεσμευτική. Νομίζω ότι εμείς τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές που το συζητήσαμε στην ομάδα μας ε, προτιμούμε να μείνουμε εδώ στην θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πιο εθελούσια μορφή και να μπορέσει ο κλάδος να αυτορυθμιστεί έτσι ώστε να αποφύγουμε απώλεια μερίδιων αγοράς που θα μπουν ε, σε αυτά οι Κινέζοι και άλλοι που έχουν άλλη δικαιοδοσία. Προφανώς αυτό θα, θα χρειαστεί ένα παγκόσμιο συντονισμό. Δεν μπορεί μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε να ε, ρυθμίζουν, που είναι και μεγάλοι ε, πλέκτες εκεί και επενδυτές. Προς το παρόν η ομάδα μου δεν υποστηρίζει αυτό που προτείνει ο κ. Μπουτικόφερ για υποχρεωτικό δεσμευτικό πλαίσιο. Προτιμούμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και συμφωνώ να αναθεωρηθεί εν καιρό, αν πραγματικά αποτύχει αυτό, όπως είπε ο κ Νάρτ, ε, Βεβαίω να αναθεωρήσουμε την κατάσταση ε, σε ένα ε, λογισμένο χρονικό διάστημα. Και υπάρχει το άλλο ερώτημα, σε ποιο βαθμό όλο αυτό θα συμπεριληφθεί στο τι τύπη θα, θα γίνει όμοιρος για να αντιμετωπίσουμε την νομοθεσία και το εμπόριο με τρίτες χώρες. Ε, δεν είναι το παρόν, στο παρόν δεν υποστηρίζουμε τις περισσότερες τροπολογίε του κ. Μπουτικόφερα από την ομάδα μα. Είμαστε υπέρ του θελοντικού σχήματο. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σόλτ είναι επίση και ο Και μετά θα παρακαλέσω του συναδέλφους να είναι πάρα πολύ σύντομοι. Και θα βάλουμε και χρονικό όριο γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει. Κανονικά αυτό το θέμα θα έπρεπε να έχει τελειώσει μέχρι τις 4.30. Ήδη είμαστε εκτό χρόνου. Beyond that limit. Thank you. So, Mr. Thank you, Mr. Ο κύριος Σόλτς, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί είχα άλλη σημαντική συνεδρίαση για το TTIP στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και έπρεπε να τρέξω να έρθω εδώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ σκληρή δουλειά. Είχαμε την ευκαιρία και σε διμερείς ε, επαφές να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Είναι από τα σημαντικότερα πιστεύω που εξετάζουμε από κοινού οι επιτροπές ΙΝΤΑ και ΑΦΕΤ. Διότι πόσοι πόλεμοι θα χρειαστούν ακόμα, πόσοι νεκροί, πόσα παιδιά να υποφέρουν από την σκλαβιά και τις ε, ε, εξωφρενικές συνθήκες εργασίας για να το πάρουμε σοβαρά υπόψη και να λάβουμε μια απόφαση στο Κοινοβούλιο. 43 κράτη του ΩΣΑ μέλη έχουν συμφωνήσει Θα πρέπει οι εταιρείε να ελέγχουν τους προμηθευτές τους και την αλυσίδα εφοδιασμού. Και θυμίζω στους αδέρφους ότι και τα 43 ε, μέλη ε, του ΩΣΑ, μεταξύ αυτών είναι και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είναι τόσο περίπλοκο να ε, ξεπεράσουμε τα εσκαμένα για να βρούμε μια λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια πρόταση που κατά την άποψή μου ε, υπολείπεται του στόχου αυτού και έχει δίκιο ο κύριος Μπιουτικόφερ, χρειάζεται αλλαγή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι για την ομάδα μου, την ΚΟΕ, θα πρέπει να είναι ε, υποχρεωτικό αυτό το σύστημα και να διευρυνθεί και το πεδίο εφαρμογή των εταιριών, δηλαδή και ακόμα και των υλικών. Ήθελα να πω ότι όταν συζητούμε για ε, μεταλλεύματα από περιοχές σύραξης, μιλούμε για μια συγκεκριμένη γεωγραφική επιρροή, ε, περιοχή συγγνώμη, και βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να το επεκτείνει αυτό και αλλού. Αλλά να δούμε και στο μέλλον τι θα γίνει. Και θα ήθελα να θυμίσω τη συζήτηση που είχαμε για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Και υπάρχουν και άλλα μεταλλεύματα από περιοχές σειράξεων που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Θα πρέπει να αλλάξει λοιπόν η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να το καταφέρουμε να πριτανεύσει η κοινή λογική στι διεπιτροπέ μα και να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Ε, πρώτον, δεσμευτικό και δεύτερον και περισσότερε εταιρείε να ενταχθούν. Ευχαριστώ. Ο κύριο Καστάλτο, μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι το να συζητούμε αυτό το θέμα σε αυτήν την Επιτροπή είναι μια τεράστια ευκαιρία να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνεκτική και υπερασπίζει τις αρχές της και τις αξίες της. Ε, βέβαια, ε, η πρόταση της Κομισιόν, ε, το να τη δεκτούμε, καθώς είναι ιδιαίτερα μινιμαλιστική, θα είναι μια χαμένη ευκαιρία, γιατί ξέρουμε ότι τους πολέμους, οι πόλεμοι δεν γίνονται χωρίς στρατιώτες και χωρίς οικονομικά συμφέροντα γι' αυτό εγώ θα αποθήσω και με ε, τροπολογίες που καταθέσουν άλλοι συνάδελφοι, ε, το να ε, έχουμε ε, μία διεύρυνση του καταλόγου των μεταλλευμάτων και να διευρύνουμε το κατάλογο για τις χώρες όπου υπάρχει κατάρρευση των οικοδομών γενικευμένη βία και επίσης θεωρώ ότι είναι σκόπιμο Αυτές οι διατάξεις πέρα από το να είναι υποχρεωτικές ε, θα πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόζονται και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Φυσικά κατανοώ ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Εδώ θα πρέπει να παρέμβουμε έτσι ώστε να υποστηρίζονται επαρκώς και να τους δοθεί και ένα σύστημα κινήτρων. Όμως δεν μπορούμε να παραμένουμε τυφλοί και κουφοί μπροστά ε, σε αυτό που ε, έχει συμβεί ε, μέσω των σειράξεων για τα μεταλλεύματα. Εγώ ελπίζω η έκθεση αυτή να μπορέσει να μπει στη σωστή οδό με την συνεργασία και με τους όλους συναδέλφους και ευχαριστώ τον εισηγήτη για το έργο του ως τώρα. Ευχαριστώ. Σας Χάουσερ για 1,5 λεπτό. Ναι κύριε Πρόεδρε. Το 2004 Ήμουν σύμβουλος του Αντιπροέδρου της, ε, του RDC, της ε, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ο οποίος είχε στο χαρτοφυλάκιό του τα μεταλλεύματα μεταξύ άλλων. Ήμουν εντολολήπτης της κυβέρνησής μου και του Υπουργείου Εξωτερικών. Τι είδα λοιπόν τότε στο Κονγκό. Είδα διαμάντια από τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό να βγαίνουν πιστοποιημένα από την κεντροαφρικανική δημοκρατία. Είδα σπάνια μέταλλα που δεν παρήγαγε η Ρουάντα να βγαίνουν από την Ρουάντα πιστοποιημένα από την κυβέρνηση της Ρουάντας και με τη στήριξη των Ευρω... μιας ευρωπαϊκής κυβέρνησης που δεν θα σας αναφέρω και με τη στήριξη μιας ε, ε, κυβέρνησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι και η πρώτη δύναμη άλλωστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, τα δίκτυα τα μαφιόζικα συνδέονται άμεσα με τις μυστικές υπηρεσίες, με τις χώρες και μάλιστα εξυπηρετούν εθνικά συμφέροντα. Και αυτό συμβαίνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να νομοθετήσουμε. Εγώ είμαι υπέρ πάρα πολύ αυστηρή τηρού περιορισμού νομοθετικού στο θέμα αυτό και πρώτο καθήκον του Κοινοβουλίου μας είναι η πληροφόρηση, η ενημέρωση. Ας φτιάξουμε ένα τμήμα πληροφόρησης και ενημέρωσης, ας προστατεύσουμε τις πηγές της ε, πληροφόρησης και όταν ανοίξει αυτό το κουτί της Πανδώρας και μάθουμε τι γίνεται στην πραγματικότητα, τότε θα έχουμε ένα κόσμο με περισσότερη και καλύτερη διαφάνεια. Ας μην υιοθετήσουμε διαδικασίες οι οποίες τελικά καθόλου δεν πλήττουν τα διάφορα κυκλώματα και τις μαφίες που κρύβονται πίσω από αυτά τα μέταλλα και μεταλλεύματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παντσέρη για ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Απλώς λίγα δευτερόλεπτα για να πω ότι υποστηρίζω πλήρως ε, τα λογικές προτάσεις του εισηγητή. Είναι επίμαχο το θέμα, όμως θα πρέπει το κοινοβούλιο αυτό να επιδείξει μια συνεκτικότητα. Στην επόμενη ολομέλη εμείς θα εγκρίνουμε την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ένα από τα κεντρικά στοιχεία της έκθεσης αυτής είναι ότι αυτό το θέμα το θεωρεί ως ένα από τις αιτήσεις για την ε, έλλειψη του σεβασμού των δικαιωμάτων. Ε, τώρα εδώ το πρόβλημα είναι ότι η ευρωπαϊκή πολιτική κινδυνεύει να μην είναι συνεπή με το τι πρέπει να κάνουμε σε εκείνη την επικράτεια. Εγώ είμαι σίγουρο ότι πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι το τέλο για να περάσουμε στον υποχρεωτικό χαρακτήρα και επιμένω και ζητώ από τον συγητή να επιμείνει στο θέμα αυτό. σα. ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάρβερ, για μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Φυσικά αναγνωρίζω τη σημασία του θέματος αυτού. Εδώ ε, βλέπουμε κάτι πολύ σοκαριστικό στην ε, Ολομέλεια. Πρόκειται για ένα ε, εμπόριο. Εμείς ε, έχουμε ήδη νόμιμη διεθνή αρχιτεκτονική, έχουμε μέτρα του ΩΣΑ και τα 28 κράτη-μέλη επίσης είναι μέλη του ΟΣΑ, τα 21 από τα 28. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς είναι ένας διαμεσολαβητής μεταξύ των διεθνών οργανισμών και των κρατών μελών. Η Κίνα συνεχίζει να είναι ένας μεγάλος καταναλωτής των μεταλλευμάτων που έχουμε σε αυτή την νομοθεσία, ιδίως στην Αφρική, όπου πολλές αντάρτικες ομάδες ε, ε, δραστηριοποιούνται σε αυτές ε, τις χώρες και σε όμορες χώρες και μάλιστα η Κίνα ε, δεν θα δεχτεί ένα σύστημα αστυνόμευσης, δεν θα λειτουργήσει αυτό. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τα διεθνή πρότυπα για την εξαγωγή και την εισαγωγή με τα τωρινά μέτρα φαίνεται ότι μια διακυβερνητική προσέγγιση είναι καλύτερη για να πετύχουμε αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε ε, διεθνή πρότυπα και να μπορούν να συμμετέχουν και χώρες ε, όπως η Κίνα. Ε, πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και ως ε, αυτό το πιστοποιητικό προέλευσης μπορεί να εκδοθεί ε, μέσω κάποιας απάτης. Έχουμε, μία, αν έχουμε μία νομοθεσία πολύ αυστηρή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε αρνητικές συνέπειες. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να λάβει και εκείνο το λόγο για 1,5 λεπτό. Ίση μεταχείριση έχουμε εδώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τι να κάνω, θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομο. Ακούσαμε την ε, πρωτοβουλία Ντότ Frank, ακούσαμε την νομοθετική δράση στο Κονγκό, τον ε, ΟΣΑ για την δέουσα επιμέλεια θα ήθελα να πω και να τονίσω ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες από μόνες τους δεν μπορούν και να αντιμετωπίσουν ε, το κακό στη ρίζα του, της βίας και της αποσταθεροποίησης. Το είδαμε, ιδιαίτερα στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Και δεν έχει καταφέρει να σπάσει ε, ο συσχετισμός αστάθειας και σειράξεων σε χώρες που έχουν τέτοια μεταλλεύματα. Γι' αυτό χρειάζεται ε, συνολική ε, αντιμετώπιση, επίλυση των διαφορών, ειρήνευση, κράτος δικαίου, αηφόρος, ε, βιώσιμη ανάπτυξη και βεβαίως διαφάνεια στην αλυσίδα ανεφοδιασμού. Γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνουν αυτά και θέλω να προειδοποιήσω η Dot Frank ε, στις χώρες των μεγάλων λιμνών και η επιρροή τους και αντίκτυπος είναι θέμα συζήτησης. Το Κοινοβούλιο έχει κάνει και αυτό έχει επιβάλει ένα de facto ε, εμπάργο ε, μετά τον Dot Frank δεν υπάρχουν ούτε αμερικανικές ούτε ευρωπαϊκές εταιρείες που να αγοράζουν από εκεί μεταλλεύματα με ολέθριες συνέπειες για ε, τους τόπιους πληθυσμούς. Στο 2014 οι εξαγωγές κασιτέρου έχουν πέσει στο μισό σε σχέση με την περίοδο 2008-2009. Ολοκληρωμένη προσέγγιση, τελειώνω, είναι αυτό που χρειάζεται και βασίζεται στην αρχή do no harm. Ε, αυτό το ξέρει η κυρία Μογκερίνη και σημαίνει εθελοντική προσέγγιση ε, όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην πληγούν οι ντόπιοι πληθυσμοί και βασιζόμενοι στον ΩΣΑ. Έχουμε ε, υποστηρίξει και περιφερειακή πρωτοβουλία για τις πιστοποιήσεις με τη Γερμανία, την αποστολή του ΟΗΕ και την κυβέρνηση του Κονγκό. Σιγά σιγά αυξάνεται 67% ε, του κασιτέρου, του βολφραμίου και του τανταλίου είναι από περιοχές χωρίς σειράξεις, ακριβώς λόγω της αυτοπιστοποίησης της τοπικής. Ε, γι' αυτό θέλουμε να προειδοποιήσουμε προσοχή, όχι υποχρεωτικές ε, ρυθμίσεις γιατί κάνουν τεράστιο κακό και στις μεγάλες λίμνες και γενικότερα στην Αφρική. Ο κύριος Μπουτικόφερ για να ολοκληρώσει σύντομα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρχίζω από το τελευταίο σημείο, αυτό που ακούσαμε τώρα. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αυτό τον κανονισμό, υποσχέθηκε ο κύριος Ντεχόχτ ότι θα φέρει ένα πιο φιλόδοξο κανονισμό από τον Ντότ Φρανκ. Και τώρα ακόμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι φτάνει, τους φτάνει το do no harm. Εμάς δεν μας αρκεί αυτό να μην βλάψουμε κανέναν εκεί πέρα. Και τους έχουν πιέσει τα λόμπι και έπιασε αυτό ορισμένες εταιρείε που δεν θέλουν να υπάρχουν αυστηρές ρυθμίσεις. Και να μην το συγκαλύπτουν και να μας λένε οι καημένοι ε, άνθρωποι που υφίστανται εκεί εκμετάλλευση να μην πάθουν τίποτα οι πληθυσμοί. Και γι' αυτό δεν θέλει η Κομισιόν ισχυρότερες ρυθμίσεις. Ε, αυτό είναι πραγματικά κρίμα ε, και θα πρέπει να το ρυθμίσουμε. Θα κοιτάξω εγώ τι θα κάνω. Εγώ πρότεινα ρυθμίσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, κάτι αξιοδότηση πράξης για να διευρυνθεί ενδεχομένω ε, το πεδίο εφαρμογή και γεωγραφικά και ως προς τα στοιχεία και τα μεταλλεύματα και κάποια άλλα στοιχεία ευελιξίας. Αλλά εάν δεν πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε από κοινού θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα πράγματα παγκοσμίω και θέλουμε μόνο να κινηθούμε αν κινηθούν και οι Κινέζοι μαζί μας, χαιρετίσματα. Τότε γιατί διαπραγματευόμαστε το TTIP. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνω τη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, σκιώδης εισηγητές, συνάντηση 26 Φεβρουαρίου, έχει προγραμματιστεί για την 9η Μαρτίου ψηφοφορία στο Στρασβούργο. Ανέβαλε, όπως ακούσαμε, ίντα τη δική της ψηφοφορία 13-14 Απριλίου και στην Ολομέλεια προβλέπεται να πάει 18 με 21 Μαΐου. Γρήγορα περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η έκθεση για την Αλβανία. Και θα παρακαλέσω τον Κνούτ Φλέκενστάιν να λάβει το λόγο. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, από τις 30 Ιανουαρίου έχετε όλοι το σχέδιο έκθεσης μου για την Αλβανία. Περί τίνος πρόκειται εδώ. Είναι μια πρώτη, ένα πρώτο σχέδιο έκθεσης ως νέος εισηγητής του νέου κοινοβουλίου για την Αλβανία την έχω εκπονήσει. Γι' αυτό αρχές ε, Ιανουαρίου πήγα στα Τύρανα, επί που είχα πολλές συνομιλίες και επαφές. Η Αλβανία τα περασμένα χρόνια έχει κάνει εντυπωσιακές μεταρρυθμίσεις και βήματα πρόοδου. Και πολύ δικαίως τον Ιούλιο του 2014 έλαβε το καθεστώς υποψήφιας χώρας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το καθεστώ τη υποψήφια χώρα είναι μια ενθάρρυνση για τι μεταρρυθμίσει που προχώρησαν και για να προχωρήσουν και να ενταθούν έτσι περαιτέρω. Ταυτόχρονα όμω είναι και μια υποχρέωση που έχει αναλάβει η κυβέρνηση τη χώρα να προχωρήσει τι μεταρρυθμίσει. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι να αποφασίζονται μεταρρυθμίσει, αλλά να υλοποιούνται επιτυχώ. Η έκθεση μου λοιπόν έχει να κάνει με τις πέντε προτεραιότητες που όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Αλβανία ε, την έδειξε υπόψη για να είναι όριμη η χώρα για την επόμενη διαδικασία, το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων για την ένταξη, που θα πρέπει να αρχίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί θα είναι ακόμα ένα νέο κίνητρο για νέες μεταρρυθμίσεις και πρόοδο. Όσο ε, ε, Βεβαίω χρειάζεται φιλόδοξη, που είναι φιλόδοξη, η μεταρρύθμιση του δημοσίου και της διοικητικής μηχανής ε, για να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα. Μια νέα νομοθεσία ε, για τη δημόσια διοίκηση έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ήδη. Η ε, Αλβανία κάνει τη δημόσια διοίκησή της τώρα επαγγελματική και την αποπολιτικοποιεί τα τα ταυτόχρονα τη διαφθορά. Όχι μόνο εγώ, δεν παίρνω μόνο εγώ δηλαδή γράμματα από πολίτε της Αλβανία για θέματα διαφθορά στη δημόσια διοίκηση. Ξέρω ότι και ο συνήγορο του πολίτη στη χώρα ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του συνήγορου του πολίτη ε, της Αλβανίας για να εφαρμοστούν στην πράξη. Και ήθελα να το πω εδώ παρουσιάζοντας την έκθεσή μου. Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα της τροποποίησης της δικαιοσύνης. Ε, για να ενταθεί και να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη της χώρας τους. Η Αλβανική Βουλή έχει συστήσει ειδική επιτροπή ad hoc για να παρακολουθεί τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης στον τομέα της δικαιοσύνης. Η έκθεση τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει επικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των ενεχομένων σε μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση. Επίσης, είναι σαφής και εδώ ε, ε, ε, υποχρέωση και της αντιπολίτευσης να συνεργαστεί, κατά πολέμηση διαφθοράς και οργανισμένου εγκλήματος. Σε όλα τα επίπεδα πρέπει να γίνει αυτό. Για να υπάρξει επιτυχία χρειάζεται συντονισμός των προσπαθειών μεταξύ όλων των θεσμών και όλων των επιπέδων. Καθώς επίσης και καλά καταρτισμένο προσωπικό. Η αλβανική κυβέρνηση πρόσφατα μας έδωσε την απόδειξη ότι είναι σε θέση να κάνει μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος και της διαφθοράς. Οι μέχρι τώρα επιτυχίες τώρα θα πρέπει να διευρυνθούν και να ε, δώσουν ε, τη θέση τους σε μια στρατηγική αντιμετώπιση και προσέγγιση. Όλα αυτά είναι σημαντικά ορόσημα στο δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνει όμως όριμη η Αλβανία έτσι ώστε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται βιώσιμες, βιώσιμες μεταρρυθμίσεις. Έχουν γίνει κάποια θετικά και κάποιες αλλαγές ας πούμε στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Αλλά αυτά θα πρέπει να είναι αισθητά για κάθε πολίτη της χώρας, στην καθημερινότητά του. Και οι βιώσιμες μεταρρυθμίσεις θα πετύχουν μόνο εφόσον όλοι οι πολιτικοί ενέχονται ε, συμμετέχουν ενεργώς. Το Δεκέμβριο πήγαμε με τον κύριο Κούκαν στην Αλβανία για να φροντίσουμε ακριβώς το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης να ξανά στο Κοινοβούλιο και να αρχίσει να συνεργάζεται. Ε, και εδώ τονίζει η έκθεση πόσο σημαντική είναι ε, επικοδομητική, πολιτική συνεργασία, διάλογος, η άμυλα για να αναζητηθούν οι καλύτερες ιδέες. Στη δημοκρατική διαδικασία το θέμα δεν είναι ε, οπωσδήποτε να έχουμε κάθε φορά συνένεση μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Αλλιώς δεν θα υπήρχε άλλη πια εναλλακτική λύση σωστή για τους εκλογείς και τους ψηφοφόρους. Το θέμα είναι να βρίσκει συμβιβασμό ε, που εκπροσωπεί καλύτερα τα συμφέροντα των πολιτών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Αυτό θα αυξήσει τελικά και την εμπιστοσύνη ε, στις δημόσιους θεσμούς και ε, σε αυτό εμείς ε, βασιζόμαστε. Είναι σημαντικό για την αλβανική κοινωνία των πολιτών να έχει ένα ισχυρότερο ρόλο στο δημοκρατικό βίο και την πολιτική ζωή της χώρας και στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης. Γι' αυτό η έκθεση καλή είναι στο εξή, το συντομότερο, και τώρα χαιρόμαστε που η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει αρχές Μαρτίου, να συνεδριάσει ε, το Εθνικό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Να αρχίσει να εργάζεται, εν πάση Αυτό το Συμβούλιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ανεξαρτήτων θεσμών, κατά κύριο λόγο, οπωσδήποτε. Αυτοί θα πρέπει ε, να έχουν αρκετό χώρο και ουσιαστική συμμετοχή. Προφανώς η έκθεση ασχολείται και με άλλα θέματα ουσιαστικά, όπως είναι οι θρησκευτικέ η ε, ε, σχέση μεταξύ εθνοτήτων, η κατάσταση των μειονοτήτων, η ελευθερία των μέσων επικοινωνίας και η σχέση καλής γειτονίας. Ακριβώς στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής και σε σχέση με τις σχέσεις με τους γείτονες, στην έκθεσή μου θα βρείτε λόγια σαφή και επενετικά. Η Αλβανία έχει αποδειχθεί επικοδομητικός γείτονας που ε, βοηθάει και συμμετέχει ενεργά στη σταθεροποίηση της περιφέρειας. Είναι αξιόπιστος εταίρος του ΝΑΤΟ και συνεργάζεται για την ε, καταπολέμηση τρομοκρατίας στην πρώτη γραμμή. Η ένταξη της ε, Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ολοκληρώνεται ούτε είναι υπόθεση μιας κυβερνητικής θητείας, μιας μόνης κυβέρνηση. Αυτή η διαδικασία δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, ανήκει στη χώρα και στο λαό της θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι η αλβανική κυβέρνηση σε όλες ε, τις προσπάθειές της υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει εθνική συνένεση για το στόχο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό η έκθεση προτείνει δυνατότητες μεγαλύτερης συμπερίληψης ε, των ε, φορέων της κοινωνίας χωρίς να λησμονεί την διακοινοβουλευτική συνεργασία. Η Αλβανία είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο χαιρόμαστε για κάθε επικοδομητικό συγκεκριμένο βήμα μεταρρύθμισης που φέρνει τη χώρα αυτή πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ χαίρομαι για την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων για τις βελτιώσεις και τις συμπληρώσεις που θα κάνουν και οι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κούκαν παρακαλώ. Και εσείς. Σας παρακαλώ να μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά, εάν μπορείτε. Οι σκιώδεις εισηγητές θα έχουν δυόμιση λεπτά και οι λοιποί θα έχουν δύο λεπτά. Όμως ο κύριος Κούκαν είναι σκιώδης εισηγητής μαζί με τον κύριο Κιούτσουκ που θα μιλήσει αργότερα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Κούκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την έλευση αυτής της έκθεσης και να συγχαρώ τον εισηγητή για την θετική και προσωπική του ε, δέσμευση, συμμετοχή στο θέμα της Αλβανίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πρέπει να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυ στην εξέλιξη της χώρας και πιστεύω ότι οι βασικές πολιτικές ομάδες μπορούν να υιοθετήσουν ε, μια κοινή στάση έναντι ε, της διαδικασίας προσέγγισης Αλβανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη γνώμη μου η έκθεση είναι αρκετά ισορροπημένη σε σχέση με τα πιο βασικά προβλήματα της χώρας και σίγουρα στη συζήτηση για τις τροπολογίες θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το κείμενο η Αλβανία έλαβε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας μετά από πολιτικές εντάσεις στη χώρα και μάλιστα Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη διαδικασία αυτή ήταν το υψηλό επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Χαίρομαι διότι η έκθεση τονίζει τη σημασία που έχει ο διάλογος στην πολιτική, η εξέβρεση συμβιβαστικών λύσεων και η βούληση να βελτιωθεί η πολιτική κουλτούρα και αυτό αφορά και τις δύο πλευρές, και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Η Αλβανία είναι μια χώρα όπου και τα δύο πολιτικά στρατόπεδα μπορούν να συνεργαστούν σε ποιο πεδίο, στο πεδίο της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η συνεργασία των δύο πολιτικών στρατοπέδων είναι αυτό που θα επιταχύνει τη διαδικασία. Άλλωστε όλο αυτό έχει σχέση και με την πολιτική κρίση που αντιμετώπιζε η χώρα. Ο πολιτικός διάλογος θα πρέπει κατά κύριο λόγο να λαμβάνει χώρα μέσα στα θεσμικά όργανα, στους θεσμούς αν θέλετε που έχουν σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό. Και θα πρέπει να ασκούμε πίεση για συμμετοχική πολιτική ε, συζήτηση, διάλογο, να αποθαρρύνουμε τον μποϊκοτάζ ε, που μπορεί κάποιος να κάνει στο κοινοβούλιο ή στις εκλογές. Ενθαρρύνουμε τους πολιτικούς μας ε, εταίρους να εργαστούν περισσότερο πάνω στις βασικές πολιτικές προτεραιότητες. Είναι καλό διότι η πλατφόρμα αυτή θα ξεκινήσει τη δουλειά της σύντομα. Το κράτος δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς του οργανωμένου εγκλήματος είναι εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα. Η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και η ανεξαρτησία αυτής είναι μία από τις προτεραιότητες. Οι σημαντικές διάφο... μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ε, η μεταρρύθμιση των ΟΤΑ. Όλα αυτά πρέπει να υπογραμμιστούν στην έκθεση. Γνωρίζω ότι Υπάρχει πολιτική αμφισβήτηση αυτών των προτινόμενων μεταρρυθμίσεων στην Αλβανία. Ελπίζω όμως ότι στην τελική θα βοηθήσουν οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα να έχει καλύτερη δημόσια διοίκηση, καλύτερους, καλύτερα στελέχη σε αυτήν, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία προσέγγισης της ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποστινάρου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω ρουμανικά τη μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα να χαιρετήσω καταρχάς τους συναδέλφους από τις δύο πολιτικές ομάδες, από το ΕΛ και τους σοσιαλιστές, που έχουν συμβάλει στο να κατευναστούν τα πνεύματα ε, στη χώρα αυτή. Τα πολιτικά πνεύματα τα οποία ήταν ιδιαίτερα οξυμένα στο παρελθόν. Και θα ήθελα να χαιρετήσω τη δέσμευση της κυβέρνησης και δεν θα πω ονόματα, ούτε θα αναφέρω για το ποιες πολιτικές ομάδες πρόκειται, θα ήθελα να χαιρετήσω την αλβανική κυβέρνηση που έχει ξεκινήσει μια διοικητική μεταρρύθμιση άνευ προηγουμένου. Αυτό είναι ένα δείγμα τεράστιου πολιτικού ε, θάρρου και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια αληθινή δημόσια διοίκηση, ουσιαστική. Και θέλω να χαιρετήσω τη θαραλέα δέσμευση της αλβανικής κυβέρνησης να καταπολεμήσει τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Εάν οι διάφορες δομές του οργανωμένου εγκλήματος μπορεί να έχουν αποφασίσει να βάλουν βόμβες δίπλα στα κτίρια όπου κατοικούν Αλβανοί αξιωματούχοι, αυτό δείχνει ότι έχουν αποσταθεροποιηθεί. Και αυτή η προσπάθεια, αυτό το τεράστιο πολιτικό θάρρος θα πρέπει να υπογραμμιστεί και από το Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ήθελα και να, να τονίσω την ουσιαστική συμβολή της Αλβανίας στην περιφερειακή συνεργασία. Η Αλβανία συνεργάζεται σε περιφερειακό επίπεδο με εξαιρετικό τρόπο, δείχνει το θάρρος της δέσμευσης της κυβέρνησης της Αλβανίας, η οποία θέλει να έχει σωστό πολιτικό διάλογο με όλες τις γειτονικέ της χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών των Βαλκανίων που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ρουμανία. Και αυτές τις προσπάθειες πρέπει να τις υπογραμμίσουμε, να τις χαιρετήσουμε και το ίδιο πρέπει να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι μπορούν να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι εφικτό δεδομένων των επιτευγμάτων της χώρας και δεδομένων των μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει. Όλα αυτά έχουν γίνει και είναι απαραίτητα για να έχει αξιοπιστία η διαδικασία ε, προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι καθήκον της, του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμβάλλουν για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και δεν θα πρέπει να δίδεται σημασία στις διάφορες, ε, ε, στους διάφορους ισχυρισμούς για ισχυρό μουσουλμανικό στοιχείο σε αυτή τη χώρα. <laughs> Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάσκου, σας ευχαριστώ και εγώ δεν είχα καταλάβει ότι τα ρουμανικά έμοιαζαν τόσο, ακούγονταν τόσο πολύ ε, όπως τα αγγλικά ή τουλάχιστον αυτά τα τελευταία που είπατε στο τέλος. Κύριε Τάνοκ για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πάσκου. Και εγώ συμφωνώ από πλευρά συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ότι πρέπει να συγχαρούμε την Αλβανία γιατί πήρε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας, είναι ήδη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Σίγουρα υπάρχουν πολλές προκλήσεις, τις αντιμετωπίζει ως μικρή χώρα γιατί είναι μικρή οικονομία, προσπαθεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, τις ε, μακροχρόνιες προβληματικές δομές και χρειάζεται μεγαλύτερη σύμπνοια μεταξύ ε, και αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι κάνουμε καλή δουλειά, ότι γίνεται σωστή δουλειά. Και κυρίως ο Πρωθυπουργός αντιράμα ότι κάνει ε, καλή δουλειά, πιστεύω. Η Αλβανία όμως είναι πλήρες μέλος του οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης και συχνά ψηφίζει en bloc ε, στο, στο αρμόδια όργανα των Ηνωμένων Εθνών για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να δούμε τι ε, ε, επιπτώσεις αυτό θα έχει το, στο μέλλον. Και πρέπει να δούμε και τι σχέση έχει αυτό με την κοινή εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφαλείας και κατά πόσο ευθυγραμμίζεται με τη δική μας. Και πρέπει να δούμε και τις ε, ε σχέσεις με τη Ρωσία ή και με άλλες χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ο τύπος θεωρεί ότι μέχρι και 500 Αλβανοί μαχητές έχουν πάει στην Συρία και στο Ιράκ και έχουν προσχωρήσει στην τρομοκρατική ομάδα ISIS. Δεν έχω καταλάβει αν είναι Αλβανοκοσοβάρι, αν είναι από την αλβανική μειονότητα ε, της Φύρωμα ή αν είναι Αλβανία από την Αλβανία. Δεν ξέρω τι πιστεύουν τα γι' αλλά ποια μέτρα υιοθετούν για να προλάβουν τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Ποια μέτρα λαμβάνουν για να μην έχουν τζιχαντιστές ε, τρομοκράτες. Ε, ποια ε, μέτρα λαμβάνουν για τη σύλληψη όλων αυτών των μαχητών εάν διαπράξουν φρικοδίες πολέμου και αυτό μπορεί να αποδειχθεί. Διότι 500 μαχητές είναι πολύ μεγάλο ποσοστό για μια χώρα 2 εκατομμυρίων κατοίκων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κιούσουκ, για μισή λεπτά. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για τις σημαντικές προσπάθειες που έκανε για να προετοιμάσει αυτή την ισορροπημένη έκθεση πρόοδου για την Αλβανία. Οι προεδρεξιακές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να οφείσουν την Αλβανία προς την επίτευξη μια εθνικής σταθερότητα είναι μια χώρα που είναι ήδη και μέλος του ΝΑΤΟ. Η Αλβανία έχει σταθερές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες. Επίσης, η εξωτερική της πολιτική ευθυγραμμίζεται πλήρως με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Επίσης, έχει υποστηρίξει τις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας πέρσι. Η Αλβανία έκανε κάποιο πρόοδο στο να σεβαστεί τα πολιτικά κριτήρια για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω περαιτέρω μεταρρυθμίσεων, η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση θα πρέπει να προβούν σε πολιτική συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Τα οικονομικά κριτήρια τώρα έχει κάνει πρόοδο για να επιτελέσει μια ε, λειτουργική οικονομία της αγοράς, πρέπει όμως να κάνει και άλλες μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πίεση. Ε, αντιμετωπίζει προκλήσεις η Ελβανία, αλλά έχει κάνει και κάποια θετικά βήματα να αντιμετωπίσει. Έχει κάνει πρόοδο κυβέρνηση στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και του δικαιοδοτικού συστήματος ε, έχει αυξήσει την λογοδοσία και τον επαγγελματισμό των δικαστών. Έχει επιδείξει η χώρα θέληση για την καταπολέμηση της διαφθοράς κατόρθωσε να βελτιώσει το θεσμικό, το θεσμικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο, το πολιτικό συντονισμό σε κεντρικό επίπεδο, όμως είναι διευρυμένη η διαφθορά σε πολλούς τομείς και στο δικαστικό σύστημα και στην εκτελεστική εξουσία και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Συμπερασματικά, ως και ο συζητητή των φιλελευθέρων, ε, θέλω να πιστήσω την προσοχή σας ε, στι ε, νομικές διατάξεις, στο είναι αρχή τη ισότητα των φύλων, στη σχετική διάταξη δηλαδή, που πρέπει να αρθεί επίσης στο ότι πρέπει να καταπολεμήσει την καταναγκαστική παιδική εργασία και να υπερασπίσει όλα τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των μειονοτήτων και να προστατεύσει και τις μειονότητες και τις υπόλοιπες ευπαθείς ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Επιτίδιος, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο εισηγητή να επενεί την κυβέρνηση της Αλβανίας για τις καλές σχέσεις που έχει δημιουργήσει με τις γειτονικές χώρες. Θα του υπενθυμίσω όμως δύο γεγονότα τα οποία δεν συνηγορούν υπέρ αυτής της απόψεως. Το πρώτο είναι ότι στην ε, Αλβανία δρούν ορισμένες πολιτικές ομάδες υπό την ανοχή της κυβερνήσεως, οι οποίες πιστεύουν στη, μεγάλη, στη δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας. Έχουν επίσημες δραστηριότητες, συγκεντρώσεις, στο, ε, στο διαδίκτυο ε, αναφέρονται και επιπλέον έχουν και σημαίες και παραστάσεις με αυτή το χάρτη της Μεγάλης Αλβανίας. Υπενθυμίζω το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη στον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων Σερβία και Αλβανία. Αυτέ οι επεκτατικέ βλέψει των ομάδων αυτών που επαναλαμβάνω γίνονται υπό την ανοχή τη ε, κυβερνήσεω τη Αλβανία έχουν επεκτατικέ βλέψει εναντίον των γειτόνων τη Σερβία, του Κωσυφοπεδίου, τη Φύρομ, τη Βουλγαρία αλλά και τη Ελλάδο. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι οπαδοί τη Μεγάλη Αλβανία διεκδικούν το εδαφικό διαμέρισμα της Υπήρου. Το δεύτερο περιστατικό που θέλω να αναφέρω είναι ότι η αλβανική κυβέρνηση καταπιέζει τα, τα ε, δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στη χώρα, κυρίως στην περιοχή της Χιμάρας, όπου δεν έχει αποδώσει τους τίτλους κυριότητος στους Έλληνες κατόχους γης. Η γη αυτή είχε δεσμευθεί από, το, από την κομμουνιστική κυβέρνηση όταν απεκατεστάθηκε η δημοκρατία και κατέπεσε αυτό το σύστημα έδωσε την γη των Ελλήνων σε Αλβανούς υπηκόους. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι Έλληνες να στερούνται της περιουσίας τους. Αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη στην έκθεσή του ο κύριος Συγητής αλλά και η Επιτροπή που ασχολείται με την έκθεση προόδου της Αλβανίας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. Preda, two minutes. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρέντα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα καταρχάς να ε, συγχαρώ τον εισηγητή για την ποιότητα του κειμένου το οποίο μας υπέβαλε. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η έκθεση αυτή πολύ εύγλωτα περιγράφει τις σημαντικές πρόοδους που έχει καταγράψει η Αλβανία το περασμένο έτος. Επίσης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο ε, πολιτική τάξη κατανόησε ε, πώς πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις. Ε, πράγμα που εμείς επανειλημμένα τονίζαμε. Βεβαίως, προφανώς υπάρχει διαφθορά και κυρίως η καταπολέμηση της διαφθοράς που παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Το υπογραμμίζει το κείμενο. Βεβαίως θα χρειαστούν επιπλέον προσπάθειες, δεν αντιλέγω. Ταυτόχρονα όμως η κατάσταση στα μέσα επικοινωνίας και η δινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Αλβανοί δημοσιογράφοι είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Και εμείς οφείλουμε να τους ε, ε, παρέχουμε την πλήρη μας υποστήριξη για να κάνουν τη δουλειά τους ανεξάρτητα. Η πολιτικοποίηση του τύπου είναι πρόβλημα. Ακόμα και αν υπάρχει αυτό και είναι πραγματικότητα στη χώρα. Επίσης πρέπει να πω ότι οι ε, πολιτικοί θύνοντες κατά στην συνάντησή μας το Δεκέμβριο έδειξαν μεγάλη οριμότητα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φαγιόν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ε, συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον εισηγητή μας για την ε, προσήλωση του και τη δέσμευση εκεί και να ε, συγχαρώ από ευκαιρία και τον κύριο Κούκαν για τα όσα ε, κατάφερε τον περασμένο Δεκέμβριο να φέρει τους πολιτικούς ε, παράγοντες εκεί ξανά πίσω στη Βουλή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί συχνά η έλλειψη πολιτικού διαλόγου χαρακτήριζε την Αλβανία και ήταν μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης θέλω ε, ως φίλη της Αλβανίας να το συγχαρώ για τη μεγάλη πρόοδο που κάνανε τους τελευταίους μήνες. Και φέτος νομίζω Υπάρχει πραγματικά αυτό το παράθυρο ευκαιρία, όπως λέγεται, για να προχωρήσει η χώρα και ειλικρινά ελπίζω οι ε, ενταξιακέ διαπραγματεύσεις να αρχίσουν το συντομότερο και να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία που έχει τώρα δημιουργηθεί. Ακούστηκαν πολλά και εγώ θα πω ότι θέλω να εθαρρύνω για να γίνουν μεγαλύτερε μεταρρυθμίσει ε, στη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, για την καταπολέμηση διαφθορά σε όλα τα επίπεδα. Ακούστηκε το θέμα του συνήγορου του πολίτη. Θα πρέπει να ε, βεβαιωθούμε ότι οι θεσμοί έχουν μεγάλη ανεξαρτησία και να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών, δηλαδή με κυβερνητικέ οργανώσει, περισσότερο στα δρόμενα και στην νομοθετική διαδικασία. Θα ήθελα επίση να πω και αυτό που είπε ένας συνάδελφος για τη ριζοσπαστικοποίηση στη χώρα είναι σημαντικό να το θέτουμε, να το συνειδητοποιούμε και να καταπολεμηθεί αυτό όχι μόνο στην Αλβανία αλλά σε όλη την περιοχή και σε όλη την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα την κατάσταση των μειονοτήτων που αναφέρθηκε, θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή για να βελτιωθεί η κατάσταση των μειονοτήτων, ιδιαίτερα να μην διακυβευθεί ε, το σύστημα ε, απαλλαγής θεώρηση διαβατηρίων για τους πολίτες. Γιατί ξέρουμε, ακούμε ότι υπάρχουν ανησυχητικά νούμερα ε, ψευδών ετούντων ασύλου που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Τζαμπάσκι. Εγώ θα ήθελα να δώσω και εγώ συγχαρητήρια στον εισηγητή. Φυσικά οι Ελβανοί έχουν κάνει μεγάλα βήματα προς τα μπρος ε, στην πρωτεξιδιακή διεκδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει η ε, Αλβανία, υπάρχει υποστήριξη από την Αλβανία της εξωτερική πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια τώρα θα ήθελα να σχολιάσω συγκεκριμένες πτυχές της έκθεσης παραδείγματο χάρη, την ανησυχία για την επιστροφή ορισμένων μαχητών. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε μία έμφαση ε, και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ θα κάνω τις σχετικές προτάσεις και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, από την Κομισιόν, ο κύριος Σαϊμον Όρντιου. Για δύο λεπτά παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ευχαριστήσω τον συγητή του κ. Φλεκενστάιν για μια καλά ισορροπημένη έκθεση πρόοδου και θα ήθελα να απηχήσω κι εγώ εκ μέρους της Κομισιόν και τις ευχαριστίες τον κύριο Κούκαν γιατί διευκόλυναν την πολιτική συμφωνία έτσι ώστε να σταματήσει τον μποϊκοτάζ της αντιπολίτευσης στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες ε, τον περασμένο Δεκέμβριο. Νομίζω τώρα ότι η ομαλή εφαρμογή αυτής της συμφωνίας είναι ζωτική σημασία ε, για να ε, υπάρχει υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στην Αλβανία. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προστατεύσουμε τις μεταρρυθμίσεις από, που σχετίζονται και προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την καθημερινή πολιτική αναταραχή. Η αντιπολίτευση έχει ε, και αυτή ευθύνη απέναντι στους Αλβανούς πολίτες με το να συνεχίσει ένα επικοδομητικό διάλογο στο Κοινοβούλιο. Τώρα, ε, σίγουρα με την χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας από το Συμβούλιο Πέρσι στην Αλβανία προωθήθηκε η διαδικασία και νομίζω ότι αναγνωρίστηκε η πρόδρος που έχει γίνει στην Αλβανία από το Συμβούλιο όμως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε και καλωσορίζουμε το γεγονό ότι το σχέδιο του κειμένου υπογραμμίζει ότι υποψήφια χώρα ότι έχει μάλλον αυτό το καθεστώς η χώρα, πρέπει να ειδωθεί ως για να ευκαιρία να της δοθεί περαιτέρω προώθηση και επίσης να κάνει περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στη δημόσια δίκη στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Και νομίζω ότι εδώ είναι πολύ καλό το ύφο στην έκθεση, καθώς τονίζεται ιδίω η ανάγκη για μια πλήρη δικαστική μεταρρύθμιση και να υπάρχει ουσιαστικά να δημιουργηθούν κάποια αρχεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να παρουσιάσουμε και θετικά τις εξελίξεις στην Αλβανία στους δικούς μας ε, πολίτες στο πλαίσιο του ε, διαλόγου υψηλού επίπεδου θα ε, προωθήθηκε μάλλον ε, η υποψηφιότητα της Λιβανίας. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε ποια είναι τα περαιτέρω βήματα που πρέπει να κάνουμε. Θέλω να αναφέρω κάτι συγκεκριμένο που έθεσε ο κύριος Τάνοκ. Συγκεκριμένα την ευθυγράμμιση της Λιβανίας ε, στις ε, θέσεις της ΚΕΠΑ. Αν δούμε τα συγκεκριμένα νούμερα, από το 2014 η Ελβενία πέτυχε 100% ευθυγράμμιση με τις θέσεις της ΚΕΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ισχυρό χαρτί της χώρας στην Ευρωπαϊκή της και μιλάμε και για δύσκολα ζητήματα όπως τη σχέση με τη Ρωσία. Επίσης θέλω να δράξω την ευκαιρία για να τονίσω από τη δική μας πλευρά ότι η θετική δέσμευση της Ελβανίας στην περιφερειακή συνεργασία επίσης εγγυάται ε, μάλλον επίσης ε, ε, εγγυάται το ότι άξια λαμβάνει τους επένους που δίνει ο κ. Φλεκεστάιν στην έκθεση. Ευχαριστώ κ. Φλεκεστάιν. Ναι, σύντομα κάποια σχόλια θα ήθελα να κάνω. Καταρχάς, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Τάνοκ, ίσως θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό το πρόβλημα των ξένων μαχητών και ιδιαίτερα ε, πώς πιο συγκεκριμένα. Από την άλλη γνωρίζω ότι ακόμα και στην Ουάσιγκτον και στο State Department ο κόσμος ανησυχεί πάρα πολύ και έχει ε, μάλλον έχει εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από τον τρόπο με τον οποίο η αλβανική κυβέρνηση ε, καταπολεμά την τρομοκρατία. Δεύτερον, ο κύριος Βρέντα είπε ότι το πρώτο θέμα εκεί δεν είναι η ελευθερία του τύπου, αλλά η ελευθερία των δημοσιογράφων και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και να κοιτάξουμε και εμείς. Τρίτον, η συνύπαρξη, η συμβίωση θρησκευτικών κοινοτήτων είναι κάτι το οποίο ε, πραγματικά ε, μπορεί να κάνει τους Αλβανούς να είναι περήφανοι γι' αυτό και μπορούν και να το εξαγάγουν όσο μπορούν προς τις υπόλοιπε χώρες γιατί είναι καλό παράδειγμα. Θα ήταν επίσης ένα καλό παράδειγμα και για την πολιτική τάξη να ακολουθήσουν αυτό. Και ένα τελευταίο για την ε, Μεγάλη Αλβανία. Αυτοί δεν παίζουν ρόλο στην πολιτική, δεν παίζουν πραγματικό ρόλο ούτε στην κοινωνία. Και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να παίξουν ρόλο ούτε στη δική μου έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα σας αναγγέλω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 3η Μαρτίου στις 6 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ και προχωρούμε στο επόμενο θέμα, στην επόμενη έκθεση πρόοδου για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και παρακαλώ τον κύριο Πρέντα να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά τον κύριο Φλέκεστάιν είναι και για μένα η πρώτη ευκαιρία που έχω να σας παρουσιάσω ε, την έκθεση πρόοδου για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Οπότε θα ήθελα να πω το εξή. Η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, κατατέθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 2014 επί κυρίου ακόμα και ήταν αρκετά ζωφερή η παρουσίαση της κατάστασης στη χώρα το 2014. Υπήρξαν μάλιστα και φωνές που έλεγαν ότι τι έκθεση πρόοδου ήταν αυτή, έκθεση μη πρόοδου είναι λέει. No progress reports σε τέτοιο βαθμό. Εγώ δεν θα το ε, έλεγα αυτό, αλλά ε, οφείλουμε να ε, διαπιστώσουμε ότι η κατάσταση είναι πιο δύσκολη στη Βοσνία ζεγοβινη από τις υπόλοιπες χώρες για τη διεύρυνση και δεν με λυπεί το γεγονός ότι ασχολούμαι εγώ με αυτή τη χώρα. Λοιπόν, να σας πούμε μερικά πράγματα για το ποιες είναι οι δυσκολίες. Κανονικά αυτό θα έπρεπε να βρίσκεται ε, στις αιτιολογικές σκέψεις του κειμένου, αλλά επειδή έχουμε περιορισμούς για τη μετάφραση, αναγκάστηκα να αφήσω στην άκρη προς το παρόν όλες τις αιτιολογικές σκέψεις. Δεν έχω βάλει καθόλου για λόγους χώρου. Και αυτά θα το αντικαταστήσω με τροπολογίες λοιπόν. Και θέλω να πω ότι η έλλειψη πολιτικής βούλησης οδήγησε σε τέλμα και οικονομικό και πολιτικό τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Η διαδικασία ένταξης ε, πλήττεται. Ε, έχει παραλύσει από την έλλειψη συνεργασίας ε, των διαφόρων μερών και υπάρχουν και εθνοκεντρικές πάρα πολλοί προσεγγίσεις. Όπως γνωρίζουμε η αρχιτεκτονική δομή της χώρας είναι πάρα πολύ περίπλοκη όσο και αναποτελεσματική και οι πολιτικοί ηγέτες δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τις μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά καθυστέρησαν σημαντικά κάθε πρόοδο της χώρας. Παραμένει η διαφθορά πάρα πολύ διαδεδομένη και κατακαιρματισμένη η δημόσια διοίκηση και υπάρχουν πάρα πολλά νομικά συστήματα που ε, είναι ανυπέρβλητα ε, εμπόδια και προκλήσεις για τη συνεργασία με την κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών που είναι και αυτοί ασθενείς. Τα δε μέσα ενημέρωσης είναι πολλωμένα και δεν έχουν ε, όλοι οι λαοί του συντάγματος, αυτό θα χαροποιήσει τους Κροάτες φίλους που αποσιάζουν κατά τα άλλα, ε, ε, έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ε, δεν εξασφαλίζονται όλα τα δικαιώματα για όλους τους πολίτες στην χώρα. Θα επανέλθω σε αυτό. Επίσης προσθέτω ότι 50% του εισοδήματος της Βοσνίας σε Ζεγοβίνη πηγαίνει στην δημόσια δίκη στα διάφορα επίπεδα. Μα είναι τεράστιο αυτό το ποσό. Τα μισά έσοδα της χώρας. Και είναι από τις τελευταίες ε, της Ευρώπης και παγκοσμίως ε, στη διευκόλυνση του εμπορίου ή στο δίκτυ ε, αίσθησης διαφθοράς. Επίσης, έχει την υψηλότερη ανεργία των νέων στην Ευρώπη, 59 παρακαλώ της 100, 15-24 ετών. 59%, 59. Όλα αυτά τι σημαίνουν. Υπάρχει μια μεγάλη δυσφορία και έχουν ξεσπάσει οι το Φεβρουάριο του 2014. Έγιναν κάποιες εκλογές τον Οκτώβριο. Δεν <coughs> πήγανε καλά, ωραία, ευχάριστα ναι αυτά, για δεύτερη συνεχή φορά, αλλά η εκλογική διαδικασία έγινε ε, χωρίς να μπορέσουν όλοι οι πολίτες να ε, είναι υποψήφοι για όλες τις θέσεις. Εγώ δεν ξέχασα το Σέιντιτς ε, Φίντσι και το λέω και στην έκθεσή μου, ξέρετε. Τέσσερις μήνες μετά τις εκλογές έχουν κάποιες προσπάθειες για τη σύσταση κυβέρνησης και του κράτους. Κανονικά 11 Μαρτίου προβλέπεται σχηματισμός κυβέρνησης. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε αυτή η ημερομηνία. Είναι η πιο αισιόδοξη εκδοχή αυτή. 11 Μαρτίου θα έχει κυβέρνηση. Έξι μήνες χρειάστηκαν μετά τις εκλογές για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Ε, είναι μεγάλη περίοδος εξαιρετικά λαμβανομένων υπόψη και των προηγουμένων. Επίσης, θα πρέπει όλοι οι θεσμοί να ολοκληρωθούν σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουν να λειτουργούν. Στην έκθεσή μου επίσης αναφέρω τα σημεία που θα πρέπει να είναι προτεραιότητες έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει προς την ένταξή της η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Βεβαίως τίθεται το θέμα τη σύσταση μηχανισμού συντονισμού, αλλιώ θα μπλοκαριστεί η διαδικασία αυτή για να μην μιλήσω για τα κοινοτικά κονδύλια. Επίσης, οι νέες αρχές θα πρέπει κατά την άποψή μου να κάνουν προτεραιότητα απόλυτη όμως την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τα είπα και στο Σαράγεβο όταν πήγα εκεί. Το έλεγα σε όλους. Τι κάνετε εσείς στα πολιτικά σας κόμματα για να πατάξετε τη διαφθορά και στους θεσμούς σας. Πολύ λίγες ήταν οι απαντήσεις. Πάρα πολύ λίγες. Ε, και γενικόλογες. Θα το ξαναρωτήσω όμως. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης έχει μεγάλη σημασία και οι μεταρρυθμίσεις και είναι προτεραιότητα. Επίσης, η ελευθερία του τύπου θα πρέπει να είναι πλήρης και εξασφαλισμένη, το λέω και στην έκθεση ξεκάθαρα. Τελειώνω, Πρόεδρε, γρήγορα. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα όσα συμφωνήθηκαν το καλοκαίρι με την Ένωση. Η ευθυγράμμισή τους με τις θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωση είναι 52% στην εξωτερική πολιτική και αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Για εμά που είμαστε τόσο πιστά μέλη της Επιτροπής μας, ευθυγράμμιση με τις θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωση μόλις 52%. Νέα προσέγγιση της Ένωση σε σχέση με τη Βοσνία είναι το πιο πρόσφατο. Είμαι σε μόνιμη επαφή με την κυρία Μογκερίνη και τον Επίτροπο Χάν του οποίου ε, συγχαίρω για τι δεσμεύσει και την προσήλωσή του, Είναι σημαντικό να παραμείνει στην εξωτερική μας πολιτική προτεραιότητα η Βοσνία. Και βεβαίως χαιρετίζω το γεγονός ότι τη γραπτή δήλωση ε, που ζητάει η νέα συμφωνία την έχουν υπογράψει όλα τα κόμματα και μάλιστα ε, αναφέρθηκε σε σημασία ιστορική κυρία Μογκερίνη. Αυτά και σταματώ I would give now the floor to... Λοιπόν, τώρα θα δώσω το λόγο στους και εισηγητές. Παρακαλώ, Παρακαλώ δυόμιση λεπτά έχετε στη διάθεσή σα. θα σας ζητήσω το σεβαστείτε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που θα παίρνουν το λόγο στη συνέχεια δύο λεπτά. Αυτό είναι το μέγιστο τη γενοδόρια που μπορώ να δείξω. Κυρία Φαγιόν. Παρακαλώ. Ο κύριο Κάν. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, επικεντρώνεται σε όλα τα βασικά όπως την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ε, αναδιάρθρωση του δικαστικού συστήματος, ε, του εκπαιδευτικού συστήματος. Ε, και ε, η έκθεση της Κομισιόν αλλά και της κοινωνίας των πολιτών κατέληξαν στο ότι δεν έχει γίνει πρόοδος και καθυστερεί σε σχέση με τους γειτονές της η Βοσνία Ριζεγοβίνη. Πάρα πολύ καιρός έχει χαθεί ενώ μεγάλωσε η δυσαρέσκεια των ε, πολιτών ε, και οι πλημμύρες στη χώρα επιδίνωσαν την ε, μιζέρια και την εξαθλίωση. Έτσι λοιπόν τώρα δίνεται μία νέα ελπίδα για τη χώρα Αυτές Οι κοινέ δεσμεύσει αυτή τη εβδομάδα είναι μία νέα ελπίδα και τώρα ανοίγει ο δρόμο για τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή καθώς η έναρξη των ε, διαπραγματεύσεων ένταξη ε, θα μπορούσε να δώσουν μια ευκαιρία στην ε, Βοσνία να προωθήσει τις μεταρρυθμίσει. Προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η επίλυση των οικονομικών ζητημάτων. Η οικονομική ευημερία βέβαια είναι μόνο δυνατή αν βασίζεται σε ένα δημοκρατικό και περιεκτικό κράτος. Παράλληλα πρέπει να συνεχιστούν και οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις, ο εκδημοκρατισμός του πολιτικού συστήματος, ε, η κατάργηση των διακρίσεων κατά των μειονοτήτων, ε, ο σεβασμός των δύο φύλων. Θα πρέπει το πολιτικό σύστημα να διασφαλίζει προσβασιμότητα σε όλους. Επίσης, δεν θα πρέπει να υποσκαπτούν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά πρέπει να προστατευτούν. Μέχρι τώρα υπάρχει μία πίεση που έρχεται από όλε τις πλευρές, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι ως νέοι πρωταγωνιστές ε, μπορούν να ζητήσουν λογοδοσία, ε, ο σχεδιασμός ε, των μεταρρυθμίσεων και εφαρμογή τους είναι ζωτική και θα πρέπει να συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών στη διαδικασία. Τα ΜΜΕ και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να ελέγχουν την κυβέρνηση, συμφωνώ, τον εισηγητή του κατά καταπολέμηση της διαφθοράς είναι απόλυτη προτεραιότητα, φύγει όλους τους τομείς, η ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών παραμένει δεσμευμένη να αποτελέσει η Βοσνία μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος Τάνοκ, δυόμιση λεπτά. Ο κύριος Τζεμπάσκι, δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για την έκθεση αυτή. Πρόκειται για την πιο δύσκολη έκθεση, καθώς ε, η κατάσταση στη χώρα αυτή είναι δύσκολο να αναλυθεί. Μιλήσαμε για την Αλβανία προηγουμένως. Αναφερθήκαμε στα ορθά παραδείγματα, όμως ε, τώρα θα ήθελα και εγώ να εκφράσω με τη σειρά μου τι ανησυχίε που εξέφρασαν και οι συνάδελφοι. Να συμφωνήσω με τι ανησυχίε που εξέφρασαν οι συνάδελφοι. Το δικαστικό σύστημα δεν λειτουργεί. Κυρίως ε, ξέρουμε ότι πρέπει να εναρμονιστούν τέσσερα ε, νομικά συστήματα. Η δημόσια δίκηση δεν λειτουργεί σωστά, είναι πάρα πολύ πολιτικοποιημένη και κατακαιρματισμένη και όπως είπα δεν λειτουργεί σωστά. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τους πρόσφυγες εντός της χώρας. Έχουμε και το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος ε, από την εποχή του φιλίου πολέμου. Υπάρχουν ε, τουλάχιστον 300 μιτζαχεντίν ε, που βρίσκονται στην επικράτεια αυτής της χώρας. Ξέρετε ότι υπάρχει και ένα βαλκανικό τάχμα εντός ενός Ισλαμικού κράτους. Δεν είναι η μόνη χώρα που έχει μουσουλμανικό πληθυσμό στα Βαλκάνια και για να αποφύγουμε κάθε απειλή θα έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί για την θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση. Φυσικά υπάρχει και το πρόβλημα τη ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση. Τα μέσα μαζική ενημέρωση δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό τι συνθήκε αυτέ. Υπάρχει και μια εθνοτική διαίρεση εντός της χώρας. Είδατε πέρσι τις διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα, ήταν κοινωνικού χαρακτήρα. Υπάρχει και πρόβλημα με την εξωτερική πολιτική σε σχέση με τη Ρωσία και η δική μας ομάδα, η ECR, θα σας παρουσιάσει κάποιες προτάσεις μέσα στις προθεσμίες που έχουν τεθεί. Σας ευχαριστώ. Κύριος Ράντος, μισή λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ θα αναφέρω δύο ακόμα ζητήματα πέρα από αυτά που αναφέρατε. Δηλαδή ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ των εθνωτικών ομάδων και υπάρχουν και πολύ χαμηλά ποσοστά επιστροφής των προσφύγων. Τι συμβαίνει δηλαδή Δηλαδή όχι μόνο νομοποιείται η εθνοκάθαρση της δεκαετίας των 90, αλλά κατά κάποιο τρόπο συνεχίζεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει έλλειψη εσωτερικών δυνάμεων. Δεν ε, ε, Θέλω να αμφισβητήσω εδώ την αντικειμενικότητα του κ. Πρέντελου. Σα παρακαλώ, δείτε την απόφαση του Συμβουλίου που αποφάσισε να εξετάσει εκ του σύνεγγυ στη Βοσνία Ριζεγοβίνη το Δεκέμβριο. Καλωσορίζω την παράγραφο 4 τη έκθεση αυτή για την ανάγκη του να συσταθεί ένα ε, μηχανισμό συντονιστικό. Πιστεύω ότι αυτά που λέγονται στην έκθεση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο μηχανισμός, ότι χωρίς αυτό το μηχανισμό θα μπλοκαριστεί η ένταξη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ε, λόγω του δυσλειτουργικού χαρακτήρα ε, του κράτους. Επομένως, είναι ζωτικό να δημιουργηθεί ένας τέτοιος συντονιστικός μηχανισμός και οι αλλαγέ στη Βοσνία Ζεγοβίνη μπορεί να έρθουν πάντοτε από τα κάτω, που είναι πάντοτε επικίνδυνο, είτε από τα πάνω. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δεσμευτούν και να αναλάβουν δράση. Αυτό που πρέπει να πετύχουμε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι η αλλαγή του συντάγματος και της δομής αυτής της χώρας διαφορετικά. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε σοβαρή αλλαγή στην πολιτική κατάσταση της χώρας. Οι συνταγματικές αλλαγές θα πρέπει να ε, δώσουν ε, μεγαλύτερη Ισχύει στους κρατικούς σφαίρους. Αυτό θα ενισχύσει τη λειτουργία του κράτους γιατί μέχρι τώρα η χώρα αυτή είναι δυσλειτουργική και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει χειρότερη κατάσταση. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε μηχανισμούς που θα προστατεύσουν τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων ε, αυτός πρέπει να είναι ο προσανατολισμός των κύριων συνταγματικών αλλαγών. Διαφορετικά θα μπορέσει να αλλάξει η κατάσταση στη Βοσνία Τζεγοβίνη. Ευχαριστώ κύριο Κόζο για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα για τη δουλειά που έκανε. Έχει μεγάλη αξία η δουλειά του και το κείμενο που προτείνει. Είναι μια πρόταση ψηφίσματος και το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι δίνει λαβή για συζήτηση επί της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βοσνία. Όμως, εδώ είναι και η παγίδα αν θέλετε, γιατί η συζήτηση αυτή δεν απεικονίζεται στο ψήφισμα. Είναι προσωρινή αν θέλετε η θέση που υιοθετεί ό,τι και να κάνουν οι Βόσνοι, ό,τι και να γίνει στην Ευρώπη. Δηλαδή ουσιαστικά υιοθετούμε προτάσεις που είναι εκτός πραγματικότητας και δεν δείχνουν ουσιαστική φιλοδοξία των ευρωπαϊκών ελίτ. Αυτό που θέλουν είναι να συνεχίσουν να έχουν μια απεικιοκρατική σχέση με τα Βαλκάνια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί επισταμένως τους νέους ηγέτες να ε, δώσουν ε, υπεύθυνε ε, λύσεις και απαντήσεις στις νόμιμες αφιβολίες και ερωτηματικά της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Και αναρωτιέμαι, γιατί να το κάνουν οι ηγέτες της Βοσνίας, ενώ δεν το κάνει καν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ηγετών της. Ουσιαστικά θέλουν οι Ευρωπαίοι με αλαζονία να κυδεμονεύσουν μια ε, πολιτική διεργασία. Υποτίθεται ότι μιλούμε για δυσλειτουργική οργάνωση της Βοσνίας λόγω διαφθοράς, λόγω οργανωμένου εγκλήματος, λόγω διαχωρισμού των εθνοτικών ομάδων και όλα αυτά υποτίθεται ότι προωθούν και τα προωθούν οι ηγέτες υπό την κυδαιμονία των Ευρωπαίων ηγετών. Οι Βόσνοι, ξέρετε, έχουν κουραστεί πάρα πολύ με όλα αυτά. Από τον περασμένο Φλεβάρι έχουμε νέα για εξεγέρσεις Βοσνίων ε, στη χώρα αυτή που δεν αντέχουν άλλο όλους αυτούς τους διχασμούς που τους επιβάλλουν και μάλιστα το λένε και στις τρεις γλώσσες και οι μαφίες που τους κυβερνούν ουσιαστικά παίρνουν εντολές από τις Βρυξέλλες και καθορίζουν τις ζωές του πολίτη από την εποχή του πολέμου μέχρι σήμερα. Αυτά που οργανώσατε πέρσι στο Σεράγεβο, στην Τούσλα, ε, νομίζετε ότι η συζήτηση ήταν για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης ή για το προενταξιακό εργαλείο όχι, ο κόσμος ζητάει ψωμί, ισότητα, ελευθερία, δημοκρατία, μέλλον και αξιοπρέπεια. Αυτό ζητούν οι Βόσνοι και αυτό θέλουν να κάνουν για να έχουν μια νέα, μια καινούργια κοινωνία. Η δημοκρατία έχει φτάσει στις ελίτ της Βοσνίας, έχει έρθει πλέον η ώρα τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλησε να καταλάβει ότι αυτοί που ήταν μέλος του προβλήματος δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης. Αυτοί που ε, ενίσχυσαν τον εθνοτικό, θρησκευτικό ή γλωσσικό πολιτικό διχασμό δεν μπορούν να συμβάλλουν στη δημοκρατία. Οι Βόσνοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για το μέλλον τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σόλτες για δύο μισή λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα, τον εισηγητή, για την πολύ καλά, η καλή δουλειά που έχει κάνει. Η έκθεση είναι εξαιρετική, είναι καλά διαρθρωμένη, είναι σαφής και ε, αντικατοπτρίζει την κατάσταση στη Βοσνία. Ωστόσο, η κατάσταση στη Βοσνία είναι πολύ ευμετάβολη και θα πρέπει η έκθεση να ενημερώνεται με νέα στοιχεία ακολουθώντας τις εξελίξεις επιτόπου. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με ό,τι ακούσαμε μέχρι αυτή τη στιγμή ως προς το κράτος δικαίου, τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Ναι, είναι η απάντησή μου. Η Βοσνία είναι μια κοινότητα στην οποία είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν αυτές οι αρχές ε, του κράτους δικαίου συμπεριλαμβανομένου και δεν πρέπει να περιμένουμε θαύματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, μπορεί να γίνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, εάν τελικά η Βοσνία αποδειχθεί ε, ως ο δράστης που ε, θα κάνει και το βήμα στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Και εκεί μπορούν να παίξει σημαντικό ρόλο και η Επιτροπή Ευρωπαϊκή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου έχει σημασία να τονίσουμε ότι η συμφωνία για το προτιμησιακό καθεστώς είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεν θέλουν να την υπογράψουν προς το παρόν και τους ασκούνται πιέσεις για αυτό το λόγο. Υπ' αυτή την έννοια οφείλουμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση ώστε αυτό να μην αποδυναμώσει περαιτέρω την οικονομία διότι ιδαλλιώς θα οπισθοδρομήσει η χώρα ακόμα περισσότερο. Η οικονομία. Η η οικονομική διάσταση της χώρας αν θέλετε σε κάθε περίπτωση είναι αυτό το οποίο θα κάνει την Βοσνία μια χώρα όπου θα ισχύσει το κράτος δικαίου όπου τελικά οι πολίτες θα πιστέψουν στους πολιτικούς τους και θα πιστέψουν στη δύναμη της χώρας τους. Ανησυχώ για το καθεστώς, ε, την κατάσταση των μειονοτήτων, την ελευθερία του τύπου, τα δικαιώματα ε, των ε, λεσβιών, ομοφιλοφίλων, φιλομεταβατικών και το καθεξής. Ανησυχώ για την ελευθερία να επικοινωνεί κανείς και κατά πόσο μπορεί μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθεξής. Υπάρχει τρόπος όμως να, ε, ε, που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να επιτύχει η Βοσνία οικονομικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο κύριος Πάσκου. Η κυρία Πετήρ για δύο λεπτά τώρα θα είναι ομιλητές, ε, θα έχουν το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, το, καλωσορίζω το ψήφισμα για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και κατά την άποψή μου ε, είναι ο δρόμος της ευρωατλαντικής ένταξης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα επηρεάσει αυτή η θετική αλλαγή της δομές. Ε, είμαι υπέρ του ευρωπαϊκού δρόμου της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, αναφανδών, για να γίνει αυτό θα πρέπει ε, όλοι οι λαοί που προβλέπει το Σύνταγμα ως συντακτικές συνιστώσεις ε, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης να έχουν ισότητα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν ένα λειτουργικό κράτος το οποίο όλοι να ε, θεωρούν ότι έχουν ίση μεταχείριση. Σήμερα αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνονται σεβαστά όλα τα δικαιώματα. Για άλλους πολίτες το κράτος είναι μητέρα, για άλλους είναι μητριά. Άρα θα πρέπει να υπάρξει πλήρης εκπροσώπηση και των Κροατών πολιτών, τα δικαιώματά τους να γίνονται σεβαστά και στο κρατήδιο της Ρεπούμπλικα Σέρψκα, αλλά και σε άλλα μέρη της Ομοσπονδίας. Έχουν όλοι το δικαίωμα να ζουν με αξιοπρέπεια και το 95% του κροατικού πληθυσμού έχουν εκδιωχθεί από κάποια μέρη και δεν τους επιτρέπουν να επιστρέψουν γιατί δεν έχουν ε, τη δυνατότητα να ε, ε, βοηθηθούν οικονομικά. Και υπάρχουν παλιές αυτόχθονες κροατικές κοινότητες που έχουν εκδιωχθεί από τις τους. Ο πολιτισμός και η θρησκεία τους έχουν καταστραφεί, η πολιτιστική κληρονομιά δηλαδή. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται στην Συρία και στο Ιράκ για παράδειγμα. Ε, ε, προστασία του περιβάλλοντος επίσης συνεχώς παραβιάζεται ο νόμος. Παράδειγμα, η συνεχιζόμενη διασυνοριακή ρήπανση Βοσνία προς Κροατία ε, από ένα δηληστήριο που υπάρχει εκεί και δεν έχει το δικαίωμα να αναπνέει καθαρό αέρα ο πληθυσμός της Κροατίας ούτε να πίνει καθαρό νερό. Υπάρχουν και διεθνείς συμφωνίες ε, που επηρεάζουν αρνητικά το βιοσύστημα του ποταμού Νερέτβα. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Πίτσουλα. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα για το ψήφισμά του, αλλά και τον τόνο που ακολουθεί στη συζήτηση. Χθε εγκρίθηκε ε, ένα κείμενο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και είναι θετικό αυτό, αλλά ήδη και τα αποτελέσματα των περσινών εκλογών θα έπρεπε να βάλουν μια κάποια πολιτική τάξη εκεί. Έχουν γίνει πολλές πρωτοβουλίες για να τερματιστεί αυτή η αποτελμάτωση στη χώρα. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τα δικά μας θεσμικά όργανα δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά θα πρέπει αντίστοιχα και οι θεσμοί της Βοσνίας να το κάνουν αυτό. Θα πρέπει εκεί οι θεσμοί να ε, εργαστούν πραγματικά στον ευρωπαϊκό δρόμο και αυτό γίνεται μόνο εφόσον υπάρξει εκεί συνένεση. Αυτά δεν επιβάλλονται ε, άνωθεν ή έξωθεν. Ε, πέρυσι, η περσινή έκθεση δηλαδή ήταν ένας κατάλογος αποτυχιών. Ευτυχώς φέτος κάπως έχει αλλάξει η κατάσταση. Καλωσορίζω ε, την παρίθμηση των διαφόρων ε, μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται οικονομικών, κοινωνικών, ενίσχυση κράτους δικαίου, καταπολέμηση της διαφθοράς που υπάρχει και σε υψηλό επίπεδο, ε, μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, να δοθεί μια όθηση για την απασχόληση των νέων και τέλος κατάργηση του ε, απαρχαιωμένου ε, συνταγματικού πλαισίου. Όλα αυτά είναι ωραία λοιπόν και εθαρρυντικά, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ο συντονισμός των προσπαθειών των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην ε, αντιμετώπιση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης που είναι και προτεραιότητα στην εξωτερική πολιτική. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη έχει πληγεί από την οικονομική κρίση που έχει προκληθεί από μια περίεργη πολιτική κατασκευή που εφευρέθηκε πριν από 20 χρόνια, αλλά ε, που έχει σπείρει όμως διχόνοια και αδικία στη χώρα. Θα ήθελα, λέει ο κύριος ε, ε Κούκα, να πω ότι είστε πολύ γενναιόδωρος πρόεδρος, κύριε Πάσκο. Δεύτερον, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την πρώτη του έκθεση για τη Βοσνία Ζεγοβίνη και ελπίζω αυτή η περίπλοκη χώρα να εξακολουθεί στο μέλλον να αποτελεί για τον ίδιο θετική πρόκληση. Τι συμβαίνει τώρα εκεί. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ την τελευταία πενταετία και παραμένω διπλωματικός στη διατύπωση. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2014 έγιναν εκλογές και μας έδωσαν ένα λόγο να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι τα πράγματα φαίνεται κάπως να κινούνται προ τα εμπρό. Η Βοσνία, η Ζεγοβίνη πραγματικά είναι πολύ ψηλή προτεραιότητα για την Ένωση. Με τη νέα προσέγγιση που έδειξαν μεταξύ άλλων η κυρία Μογκερίνη ε, μόλις χθες επισκέφθηκε τη χώρα για δεύτερη φορά και πριν από τρεις μήνες δηλαδή είχε ξαναπάει με τον κύριο Χάν είναι καλό που γίνονται, συστήνονται οι πολιτικοί θεσμοί και τώρα έχει έρθει η ώρα, η στιγμή για τους πολιτικούς ηγέτες ε, να ανανεώσουν το κοινωνικό συμβόλαιο με την κοινωνία. Τα ε, περίπλοκα προβλήματα ζητούν περίπλοκες λύσεις και λύσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του κάθε προβλήματος κάθε φορά. Τα κοινωνικο-οικονομικά κυριαρχούν ε, στην νέα προσέγγιση. Ε, και το επόμενο που περιμένουμε είναι να εφαρμοστεί πλήρω η Συμφωνία Εταιρικής ε, Μανοσύνδεσης και Σταθεροποίησης ε, και δεν θα πρέπει να το λησμονούμε. Γενικά έχω να κάνω μια παρατήρηση στο τέλος, ότι θα πρέπει να προσβλέπουμε σε θετική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία Ριζαγοβίνη. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει τώρα μια συναστρία ε, για ε, τη νέα ε, όθηση που πρέπει να δοθεί για τη χώρα. Οι πολίτες της έχουν περιμένει πάρα πολύ καιρό, υπερβολικά μεγάλο διάστημα. Ευχαριστώ η κυρία Φαγιόν. Δύο λεπτό. Um, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή. Πολλά υπόθηκαν ακούστηκαν κριτικές, αλλά φυσικά υπάρχει και καλή βούληση όλων των συναδέλφων και των συγητή να βοηθήσουν τη στην Ερσεγοβίνη. Πάντως θέλω να παραμείνω αισιόδοξη για αυτά τα δύο λεπτά, Κυρίω ε, μετά από ε, πάρα πολύ σύγχυση και απογοήτευση που ήρθε από τη χώρα λόγω της έλλειψης ε, πρόοδου και αξιοπιστίας. Χτες αυτό που συνέβησε στην Βοσνία εγώ το θεωρώ ιστορική ευκαιρία για τη χώρα. Έτσι λοιπόν αυτά τα νέα είναι πάρα πολύ σημαντικά κυρίω για του πολίτες. Μια γραπτή δέσμευση της Προεδρίας της Βοσνίας Ζεγοβίνης να προβεί στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια της διαδικασίας προσχώρησης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω πράγματι οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να συνεχίσουν λαμβάνοντας συγκεκριμένα βήματα, κάνοντας συγκεκριμένα βήματα. Δεν θέλουμε να δούμε πολιτικά λάθη του παρελθόντος. Ξέρω ότι δεν θα είναι ε, στρώμενος μοροδοπέταλα ο δρόμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά η Βοσνία Τζεγοβίνη μπορεί και πρέπει να συνεχίσει και θα πρέπει και εμείς να βάλουμε τη δυνατά μας για να τη βοηθήσουμε. Ευχαριστώ κύριο Πρέντα για συμπεράσματα. Πολύ σύντομα, γιατί δεν συμμερίζομαι 100% την αισιοδοξία της κυρίας Φαγιών. Όχι ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά μερικές φορές χάνουμε και κάποιες ευκαιρίες. Και εγώ ελπίζω ότι θα κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα η πολιτική διαδικασία στη Βοσνία. Τώρα, θα ήθελα να πω στην αντίθεσή μου σε αυτό που είπε ο συνάδελφος Περμόη σε σχέση με τη μαφία, την τοπική μαφία, παραθέτω, που υποστηρίζεται από τις Βρυξέλλες και τη Ρουάσικτον. Θα ήθελα να φυστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι Βρυξέλλες είστε κι εσείς ως μέλος του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μάλιστα ακριβώς είπατε, όπως ε, και οι άλλοι συνάδελφοι, τοποθετήκατε κατά αυτής της ντόπιας μαφίας. Τώρα, συμφωνώ με την προοπτική του κ. Σόλτες ε, που είπε ότι δεν είναι δυνατά τα θαύματα. Πράγματι. Πιστεύω ότι αυτό που περιμένουμε από τη Βοσνία είναι προσπάθειες και όχι αυτοί να αναμένουν να γίνουν θαύματα. Δηλαδή εδώ τώρα βρισκόμαστε στο επίκεντρο του προβλήματος, θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά γιατί χρειάστηκαν 6 μήνες για τη διαπραγμάτευση και πάνω από δύο εβδομάδες για να πούνε ότι συμφωνούν με τη γραπτή δέσμευση. Είναι τεράστιο το χρονικό διάστημα. Τώρα ζούμε στον 21ο αιώνα, όχι στο 18ο. Δηλαδή στις πολιτικές διαδικασίες ε, ακολουθούμε ταχύτερου ρυθμούς. Τώρα, θέλω να αναφερθώ στις συνταγματικές αλλαγές, στις οποίες αναφερθήκαν τρεις συνάδελφοι, Ράντος, Πίτλο κτλ οι συνταγματικές ε, αλλαγές ίσως ε, να έρθουν αργότερα. Εγώ θεωρώ ότι τώρα δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα συνταγματικών αλλαγών. Δεν αποκλείω βέβαια δυνατότητα ε, κάποιες πολιτικές πράξεις ε, μαζί και με τη βοήθεια κάποιων κρατών μελών και δεν είναι η πρώτη φορά, να μπορούσαν να το εξετάσουν αυτό, δηλαδή να δώσουν μια όθηση προς τις συνταγματικές αλλαγές να πιέσουν προς συνταγματικές αλλαγές. Όμως ε, εγώ νομίζω ότι τώρα δεν είναι κατάλληλη χρονική στιγμή για να γίνουν τέτοιε συζητήσεις για συνταγματικές αλλαγές. Πόσο μάλλον, για να αναφερθώ στο όσο είπε και ο κύριος Κούκαν, ε, είμαστε περισσότερο σε μια λογική της ανανέωσης του κοινωνικού συμβολέου. και να σας πω ε, και κάτι ε, που λένε ο ότι δεν ε, είμαστε τώρα ξεμολυμένοι στη φύση για να βρούμε τον γεμόνα μας. Και η τροποποίηση του χρόνου δεν είναι προτεραιότητα τώρα. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που να στοχεύουν στην ευημερία των πολιτών και στο πλαίσιο αυτό εγώ κατάλαβα την αναφορά του κύριου Κούκαν στο κοινωνικό συμβόλαιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και φυσικά με πολύ ενδιαφέρον περιμένω τις τοπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Πριν να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, κυρίως ε, Σάιμον, ότι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θέλει το λόγο. Ναι, δύο λόγια θα πω μόνο κύριε Πρόεδρε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Όπως και με τις προηγούμενες εκθέσεις θα ήθελα να συγχαίρω και για αυτήν τον εισηγητή κύριο Πρέντα. Θέλω όμως να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να σας ενημερώσω για κάτι ε, για το εξής. Μετά τις χθεσινές εξελίξεις μπορούμε να έχουμε ένα επόμενο στάδιο στις σχέσεις Βοσνίας, Βοσνίας-Ατσεγοβίνης και ΕΕ χθες το κοινοβούλιο τους υιοθέτησε τη γραπτή δέσμευση και αυτό είναι βασικό για να ανοίξει ο δρόμος για την προσέγγιση της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ελπίδα που δίδεται στους Βόσνιους πολίτες ότι μπορούν να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να πετύχουν τις φιλοδοξίες τους και ίσως του χρόνου να μην χρειαστεί να μιλήσουμε για μια έκθεση προόδου όπου γίνεται αγώνας να συμφιλειωθεί ο τίτλος της έκθεσης με το περιεχόμενο αλλά να έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα επενεί την πρόοδο που θα έχει πραγματικά ε, σημειωθεί. Ε, βασικό μήνυμα λοιπόν είναι ε, αυτό το μήνυμα που εξέπεμψε η κυρία Μογκερίνη στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας Ερσεγοβίνης, ότι δηλαδή είναι σημαντική η προσέγγιση και με βάση τα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου του 2014 το επόμενο στάδιο είναι το εξής το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποφασίσει για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Σταθεροποίησης Σύνδεσης Βοσνίας Ερζεγοβίνης μετά, 7 χρόνια μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Και άρα έχουμε εργαλείο να ε, απελευθερώσουμε τις δυνάμεις έλξης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα αυτή και μπορεί να γίνει πολιτικός διάλογος σε, υπουργικό, επίπεδο γιατί θα υπάρξει συμβούλιο υπουργικό που θα ασχολείται με την εφαρμογή της Συμφωνίας σταθεροποίηση και Σύνδεσης. Αυτό λοιπόν θα είναι το επόμενο βήμα από πλευρά Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να στηρίξουμε τις αρχές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στις πολύ σοβαρές ε, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή. Π.χ ανεργία των νέων έχει ένα νούμερο πραγματικά τρομακτικό. Ε, πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με ε, όλους τους διεθνούς φορείς, τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς μεταξύ άλλων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια σωστή δυναμική σε αυτή την πορεία, σε αυτή την κατεύθυνση της προσέγγισης δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από μια εξαιρετικά αρνητική έκθεση προόδρου ε, έχουμε δει πολλές θετικές εξελίξεις τις τελευταίες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Καταληκτική προθεσμία ε, για την υποβολή τροπολογιών 5 Μαρτίου το μεσημέρι στις 12. Τελευταίο σημείο στην ημερήσια μας διάταξη τώρα. Αναστολή της εφαρμογής τη διαδικασία σταθεροποίησης ε, και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων για χώρε και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη σχετική διαδικασία όσον αφορά βέβαια τη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Κύριε Πρέντα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καθησυχάσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που αναφέρατε το έχουμε ήδη συμπεριλάβει στην έκθεσή μας. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα αυτό, η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουνίου του 2014 είναι στην τελική αρκετά απλή, διότι στόχος της είναι να τροποποιήσει τον κανονισμό 12-15 του 2009 με εμπορικές προτιμήσεις αυτόνομες σε σχέση με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ε, που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες σύνδεσης και θα επεκταθούν οι προτιμήσεις οι εμπειρικές σε τρία επίπεδα. Πρώτον, μέχρι το Δεκέμβριο του 2020. Ε, αυτή η πρόταση έτυχε θερμής υποδοχή σε σχέση με τις δημορίες συμφωνίες με τις χώρες αυτές. Στη, υπάρχει στήριξη της ένταξης στην Ένωση και είναι σημαντικό στοιχείο όλα αυτά τα μέτρα τα προτιμησιακά για πολιτική σταθερότητα και οικονομική πρόοδο των περιοχών αυτών. Άλλωστε στην τελική ο σκοπός μας είναι αυτές οι χώρες να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα επιτρέπει να ανασταλούν αυτά το προτιμησιακό προτιμησιακό καθεστώς όταν διαπιστώνονται παραβιάσεις καταστρατηγήσεις δημοκρατίας κράτους δικαίου, δικαιωμάτων ανθρώπου και ούτω καθεξής. Αναστολή λοιπόν τέτοιου είδους εμπορικών προστιμίζων για τη Βοσνία Ερσεγοβίνη εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος της χρονιάς για την προσαρμογή της ενδιάμεση συμφωνίας σε σχέση και με την προσχώρηση της Κροατίας. Εγώ ασχολήθηκα λοιπόν από όλα αυτά, ασχολήθηκα μόνο με αυτά που άπτονται της αρμοδιότητας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχουμε την τροπολογία για την νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ξεκινήσει δηλαδή τη Συμφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης με το Κοσφοπέδιο και παρουσιάζω άλλες δύο τροπολογίες για τη διατύπωση της ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρώ ότι μια ρήτρα για ανθρώπινα δικαιώματα όταν διατυπώνεται αποφατικά δηλαδή να, να απόσχει η χώρα από την καταστρατήση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό δεν είναι ενδεδειγμένη διατύπωση θα πρέπει να έχουμε θετική, καταφατική διατύπωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και για τις αρχές του κράτους δικαίου, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις αρχές της ΚΟΠΕΧΑΓΙΣ. Δεν θέλουμε οι χώρες αυτές να σέβονται στο περίπου τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου. Δεν θέλουμε να υπάρχουν διαχωρισμοί και βαθμίδες σεβασμού, βαθμίδες και διαβαθμίσεις αυτού το οποίο, το οποίο μπορεί να γίνει ανεκτό ως παραβίαση ή καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η μόνη δυνατότητα μιας χώρας να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως ε, προτείνω τη διατύπωση που είχε χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχο εργαλείο νομοθετικό σε σχέση με την Ουκρανία που είχε εμφανιστεί και δημοσιοποιηθεί τον περασμένο φθινόπωρο και δεν βλέπω γιατί για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα έπρεπε να υιοθετήσουμε διαφορετική ε, ε, προσέγγιση. Δεν βλέπω γιατί για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να δίνουμε ε, ε, προτιμησιακές εμπορικές δυνατότητες με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το κάνουμε στο Πακιστάν και γιατί η Ουκρανία να μην μπορεί να ε, απολαμβάνει του ίδιου καθεστώτος. Ε, συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περισσότερη συνοχή, περισσότερη διαφάνεια του τρόπου με τον οποίο η παραπομπή στα ανθρώπινα δικαιώματα εμφανίζεται στα νομοθετικά κείμενα που έχουν να κάνουν με προτιμησιακό εμπορικό καθεστώ. Π.χ. θα μπορούσαν όλα αυτά να γίνουν και μετά την υλοποίηση σχετική μελέτη. Και δύο παρατηρήσει πιο γενικέ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, ω προ την αναστολή εμπορικών προτιμήσεων, εμπορικού προτιμησιακού καθεστώτο με τη Βοσνία ε, δεν χαίρομαι καθόλου με αυτή την προοπτική της αναστολής του καθεστώτος αυτού του. Ελπίζω να βρεθεί λύση μέχρι το τέλος της χρονιάς ε, ε, και χάρη στη νέα προσέγγιση της ΕΕ ως προς τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση και δεύτερον ως προς το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό. Οι δικές μας προτιμήσεις, οι προτεραιότητες πρέπει να τύχουν απόλυτου σεβασμού ως προς την απόφαση για την αναστολή των εμπορικών προτιμήσεων. Είχα εξαιρετική συνεργασία και διάλογο με τους αντίστοιχους συναδέλφους από τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ο εισηγητής ζήτησε την ε, ε, ένταξη νομοθετικής πράξης κατά εξουσιοδότηση. Ε, να υπάρξει αυτή η αναφορά στο κείμενο. Ο εισηγητής κύριος Μπετίνη, αρμόδιος επί της ουσίας. Ευχαριστώ. Ναι, Έχουμε, λέει ο κύριος Πάσκου, και τον κύριο Μπετίνη και κάποιον από τους σοσιαλιστές. Κύριε Μπετίνη, έχετε το λόγο παρακαλώ. Είναι εδώ. Τι Να ακούτε κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα συμμετοχής στη συζήτηση στην γνωμοδότηση του κυρίου Πρέντα. Εγώ παρουσίασα την έκθεση στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, μία έκθεση σχετική με την παρουσίαση από την πλευρά της Κομισιόν, μία τροποποίησης του κανονισμού του 2009. Δεν ε, θα αναφέρω τώρα όλα τα θέματα, τα αναφέρω ο κύριος Πρέντα. Εγώ συμφωνώ με το πνεύμα της έκθεσης του κυρίου Πρέντα. Υπογραμμίζω δύο πτυχές στην έκθεσή μου. Η πρώτη αφορά τα εμπορικά, τα συγκεκριμένα εμπορικά μέτρα, εγώ πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν, δηλαδή το θέμα της αναστολής την 1η Ιανουαρίου 2016 των εμπορικών προτιμήσεων για τη Βοσνία, αν δεν βρεθεί μια συμφωνία, αν δεν υπάρξει μια ε, τροποποίηση, ε, λόγω του γεγονότος ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κροατία, ε, τότε αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να λάβει χώρα αυτή η αναστολή. Εγώ εύχομαι ολόψυχα αντίθετα να βρεθεί μια συμφωνία και η ουσία αυτή τη συμφωνία θα πρέπει να είναι ότι τίποτα δεν πρέπει να αλλάξει για τη Βοσνία σε ό,τι αφορά στις εμπορικές ανταλλαγές παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να φτάσει τις εμπορικές ε, συναλλαγές που έχουμε σήμερα μεταξύ Βοσνίας Ευζεγοβίνης Ευρωπαϊκής Ένωσης να φτάσει στο επίπεδο που υπήρχε πριν από την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα παραδοσιακά προϊόντα, με τις, παραδοσιακές συναλλαγές. Εγώ πιστεύω ότι εμείς πρέπει αυτή τη συζήτηση για τα εμπορικά θέματα να την εντάξουμε σε μια πολιτική καινοτομία. Δηλαδή ότι για πρώτη φορά η Βοσνία και χάρη στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πράγματι βαδίζει ε, σε ένα δρόμο ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά εγώ πιστεύω ότι για πρώτη φορά Είχαμε μια ιστορική πράξη, δηλαδή ότι εγκρίθηκε στο Βασιλιακό Κοινοβούλιο ένα εγγραφό που προσυπογράφει από τους πολιτικούς ηγέτες και το οποίο δέχεται να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις, δέχεται τις αρχές και τις αξίες και τις δοκιμασίες που είναι απαραίτητες ε, για την επίτευξη αυτής της πορείας. Ε, υπάρχει λοιπόν μια καινοτομία γιατί έχει αλλάξει και η δική μας ε, προσέγγιση. Εμείς ε, τώρα κάπως αντιστρέψαμε τα πράγματα. Δεν ζητήσαμε από τη Βοσνία τα πιο δύσκολα, αλλά αντίθετα προκειμένου να αρχίσει να κάνει κάτι συγκεκριμένο, τη ζητήσαμε να ξεκινήσει από μικρά δυνατά βήματα. Και αυτές ήδη αυτά παγιώθηκαν από μια πράξη πολιτικής βούλησης πολύ σημαντική. Και η Βοσνία δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει μόνη της, χρειάζεται βοήθεια. Και αυτή η βοήθεια τι χρειάζεται για να ξανασηκωθεί και για να μπορέσει να λύσει τα μεγάλα προβλήματα τα οποία ανέφεραν όλοι. Και στη βοήθεια μόνο από εμά μπορεί να έρθει. Η Ευρώπη έχει και ένα συμφέρον εδώ εμείς. Έχουμε πάρα πολλά μέτωπα ω Ευρώπη. Έχουμε το μέτωπο της Ουκρανία, τη Λιβύης, έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Ε, επί των οποίων ε, πρέπει ε, να εργαστούμε για να λύσουμε γιγάντια προβλήματα. Εγώ δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε και στα Βαλκάνια μια δυσάρεστη κατάσταση, μια έρηδα και που θα μπορούσε να έχει δυσάρεστες εξελίξεις. Βασίζομαι λοιπόν στην έκθεσή μου σε αυτή την ισορροπία φενός στα εμπορικά μέτρα και στο ουσιαστικό περιεχόμενο και οθώ τη Βοσνία στο να σκεφτεί ότι οι κανόνες είναι ίδιοι για όλους και ότι δεν ε, μπορεί να υπάρχει κάποια εξέλιξη, αν δεν υπάρχει η ίδια προσαρμογή που έχουν επιδείξει και άλλες χώρες των Βαλκανίων. Όμως αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί κύρωση, αλλά ως μια όθηση προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή της ευρωπαϊκής προοπτικής. Και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις συμφωνεί και το 80% των πολιτών στη Βοσνία. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω ότι οι Βόσνοι πολίτες βλέπουν την Ευρώπη ως ε, την Ευρώπη της πλουτοκρατίας ε, που είναι έτοιμοι να τους φαγιάσουν. Αλλά έχουν και αυτοί μια ελπίδα ότι μπορούν να αποτελέσουν μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας προκειμένου να μπορέσει να είναι και το μέλλον τους ε, βιώσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τζαμπάσκι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω στο χρόνο που μου δίνεται να εκφράσω την αντίθεση της ομάδας μου. Η Βοσνία Τζεγοβίνη πολύ γρήγορα επικύρωσε τη συμφωνία για τις εμπορικές προτιμήσεις, κυρίως μετά την ένταξη της Κροατίας. Ε, με ενημέρωσαν ότι στην Επιτροπή ΙΝΤΑ η πλειοψηφία των μελών προτιμά να εφαρμοστεί η ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έτσι όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς ξεκινάμε από την ιδέα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ενισχυμένε αρμοδιότητες ε, σε ό,τι αφορά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά ήθελα να πω. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ράντο. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι Χαιρετίζω την επέκταση των ε, προτιμησιακών ε, σχέσεων με τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το βλέπουμε ε, πόσο θα βοηθήσει στην παρούσα περίοδο κρίσης για την οικονομική τους βιωσιμότητα και την πορεία τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, λυπούμε που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακολουθεί το ίδιο καθεστώς για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και χρειάστηκε να υπάρξει μια διάμεση συμφωνία. Ελπίζω ε, να ε, λάβει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Ένωση όλες αυτές τις θετικές εξελίξεις και να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αλλαγής της κατάστασης. για να μην υπάρξει αναστολή του συστήματος ε, ε, εμπορικών προτιμήσεων από την 1η Πρώτου του 2016. Εμείς πιστεύουμε και θέλουμε η Βοσνία Ριζεγοβίνη να ε, προχωρήσει και στην εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης. Ελπίζω όλα αυτά να γίνουν το συντομότερο κατά τη διάρκεια του 2015 για να μην διακοπεί η ρύθμιση αυτή. Ε, ακούσαμε, σε προηγούμενη μάλλον έκδοση έλεγε το έγγραφο ότι ε, θα αναστέλλονται αυτές οι ρήτρες σε ε, περίπτωση συστηματικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κανόνων της δημοκρατίας. Τώρα οι χώρες της περιοχής έχουν ε, αναπτυχθεί αρκετά και ε, το αλλάξαμε αυτό ως διατύπωση και λέμε ότι αναμένουμε ότι θα τηρήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα αντί να λέμε ότι θα τους τιμωρήσουμε αν δεν τα τηρήσουν. Ο κύριος Χάν, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τον, για την πρόταση και τον κύριο Πρέντα για την γνωμοδότηση. Οι σοσιαλιστές και δημοκράτες καλωσορίζουν ε, την ε, επέκταση στα Δυτικά Βαλκάνια αυτής της Ρύθμιση και αυτό συνεισφέρει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Θα πρέπει να ειδωθούν αυτά τα μέτρα στο ευρύσιο πλαίσιο των σχέσεών μας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Έκλεισε το μικρόφωνο του μιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτά τα μέτρα, έλεγα, λοιπόν, θα πρέπει να δοθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικών μας για τη σχέση των Δυτικών Βαλκανίων. Απότερο στόχος μας είναι η πλήρης ένταξη όλων των χωρών της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να προσθεθεί μια ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήταν πάγιο αίτημα αυτό δικό μας και καλωσορίζουμε πάρα πολύ αυτό τα κράτη που θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της Κοπεθάγης Και είναι σημαντικό να ενταχθεί μια ρήτρα που να εξασφαλίζει τη δράση που μπορεί να αναλυφθεί σε περίπτωση σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των θεμελιωδών ελευθεριών, κράτους δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ υποστηρίζω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υιοθετηθεί η διατύπωση GSP Plus ε, για βασικές ε, αρχές που συμπεριλαμβάνουν και ε, τα πρότυπα στα εργασιακά αλλά και τα περιβαλλοντικά κατά την άποψή μου για να προστατεύονται και να προωθούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αρχές της αηφόρου ανάπτυξης υποστηρίζω ότι ρήτρα για τη Βοσνία γιατί αναλαμβάνει δράση για την προστασία της Κροατίας που ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να υφίσταται διακρίσεις. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει ευθύνη και απέναντι στην ε, ασφάλεια και τη σταθερότητα της Βοσνίας και Ζεγοβίνης. Γι' αυτό προτείνω σε περίπτωση που έχουμε ε, οποιασδήποτε απρόβλεπτες και σοβαρές καταστάσεις να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα και αναλόγως οι Υπουργοί Εξωτερικών μας να διακοπεί η συμφωνία για να διατηρηθεί η ασφάλεια και ε, η ε, σταθερότητα στην περιοχή. Πάντως προσβλέπω στη νέα κυβέρνηση ε, της Βοσνίας Σεζεγοβίνης για να επιλύσει και τα υπόλοιπα εκκρεμή ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πιτσούλα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το σύστημα των προτιμήσεων είναι πάρα πολύ εποφελές για τις χώρες ε, των Δυτικών ε, Βαλκανίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το βλέπουμε και στην έκθεση που λέγεται ότι το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο υπαριθμόν ένα εμπορικό εταίρος οι εξαγωγές ήταν 72,2% ενώ οι εισαγωγέ 82%. Δηλαδή και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ε, αυτές οι προτιμήσεις ε, υποστηρίζουν και την περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτρέπουν βελτίωση και στο, για το πολιτικό κλίμα και την σταθερότητα όλης της περιοχής. Όταν μιλούμε για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την αδυναμία της να ενταχθεί πλήρως στην ε, εμπορική πρακτική και να ευθυγραμμιστεί με τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Τι εννοούμε. Ότι αυτό ε, θα έχει ως αποτέλεσμα ε, απώλειας ε, τριών εκατομμυρίων ευρώ μόλις. Δηλαδή είναι συμβολικού χαρακτήρα, δεν είναι μεγάλο οικονομικό ποσό. Είναι πολιτικό το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται ε, το νόμο και είναι γνωστοί οι κανόνες του παιχνιδιού από την αρχή και θα πρέπει να τηρούνται. Όταν η Ουγγαρία και η Σλοβενία ε, βγήκαν ε, από τη ΣΕΦΤΑ βρέθηκε ε, στην ίδια κατάσταση η Κροατία με τη σημερινή της Βοσνίας και χρειάστηκαν δύο γύροι διαπραγματεύσεων για να ρυθμίσουν τα θέματα ε, των σχέσεών μας με τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Ελπίζω να βοηθήσουν οι νέες αρχές προς την κατεύθυνση αυτή. Και εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πάλι ο κύριος Σάιμον Μόλτσιο. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να, καν, να ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο νομίζω είναι σημαντικό. Δεν ζητούμε από τη Βοσνία νέες εμπορικές παραχωρήσεις, ούτε περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς τους. Σκοπός του κανονισμού είναι να διατηρήσει το εμπορικό πρότυπο που έχουμε φτιάξει με τη Βοσνία και που υπήρχε πριν την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι αμφότερες πλευρές να ε, προσαρμόσουν τις ποσοστώσεις σε σχέση με τα αδασμολόγητα. Ο κύριος Πιτούλο, Πιτσούλα, με συγχωρείτε, ε, μας παρέθεσε τις συνέπειες που θα είχε κάτι τέτοιο εάν δεν είχαν διατηρηθεί εμπορικές παραχωρήσεις έγινε λόγος για απώλεια τριών εκατομμυρίων ευρώ από πλευράς Βοσνίας. Η μέγιστη εθνική απώλεια είναι αυτό το νούμερο και συμφωνούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό το νούμερο. Ας δούμε όμως και τον αρνητικό αντίκτυπο αν αρνηθεί η Βοσνία να ε, ε, ε να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσει των Κροατών εξαγωγέων οι οποίοι χάνουν 70 εκατομμύρια ευρώ ετησίω αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και η Βοσνία και όλες οι άλλες χώρες των Δυτικών ε, Βαλκανίων ευθυγραμμίζονται με αυτό. Και να σας πω δύο λόγια για τη ρήτρα αναστολής. Δεν θέλουμε να αναστείλουμε τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα. Δεν είναι η προτιμόμενη επιλογή μας αυτή. Ε, ο σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η δοκιμασμένη μεθοδολογία που ακολουθούμε τόσα χρόνια με επιτυχία ισχύει και λειτουργεί και σε αυτή την περίπτωση. Ουσιαστικά λειτουργεί ως μόχλευση, ως αντίδαρο Δηλαδή να ξέρει η Βοσνία ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς έχει την προθεσμία, τη δυνατότητα για να παρατείνει, να επεκτείνει την ρύθμιση, να προσαρμόσει τα ποσοστώσεις για τα δασμαλόγητα ή ο, ο κανονισμός από τον οποίο εποφελούνται θα πάψει να ισχύει. Και θα ήθελα να τονίσω και άλλα ε, δύο θέματα. Ως προς τη ρήτρα για ανθρωπίνα δικαιωμάτων. Ακολουθούμε τη πεπατημένη που υιοθετούν οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου σε όλα τα κείμενα που συνάπτουν με τις τρίτες χώρες. Νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσετε με τους συναδέλφους σας στην αντίστοιχη επιτροπή. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, ως προς ε, την πρόταση να εμπλακεί το Συμβούλιο σε αυτές τις διαβουλεύσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν βλέπουμε γιατί αυτό θα είχε προστιθέμενη αξία, διότι η αναστολή είναι αυτόνομη, ε, γίνεται αυτομάτως και δεν ισχύει πριν από τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας 31 12 31-12-15 και άλλωστε έτσι καθησυχάζονται οι διάφοροι ότι πράγματι θα αναστολεί η αναστολή. Θα μπορέσει να ανασταλεί η αναστολή, να αποσυρθεί η αναστολή, αναστολή αυτή όταν τα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Όσοι έχουν υποβάλει αυτή την τροπολογία ενδεχομένω θέλουν να αποφύγουν κάτι τέτοιο. Ενθαρρύνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην ψηφίσει αυτή την τροπολογία και ευχαρίστω σα το αναλύουμε και περαιτέρω και εκτό αιθούση. Ευχαριστώ ο κύριος Πρέντα για να κάνει κάποιε καταληκτικέ παρατηρήσει στη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν έχω πολλά να προσθέσω. Πολύ καλό αυτό λέει ο Πρόεδρος. Να ευχαριστήσω μόνο τους συναδέλφους λέει ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ. Κλείνουμε λοιπόν τη συνεδρίαση ανακοινώνοντας ότι στις 9 Μαρτίου θα ψηφίσουμε την, ε, το κείμενο αυτό και με αυτά και με αυτά τελειώνουμε τρία λεπτά πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Ευχαριστώ.